We will make a start. Depleted though our numbers may be. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ενδεχομένως να μην είμαστε αρκετοί ακόμα στην αίθουσα. Εγώ πάντως στις 2 και 29 μπήκα στην αίθουσα αυτή και είναι προγραμματισμένη για τις 2 και 30 η συνεδρίασή μας. Επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε, τουλάχιστον οι αντιπρόεδροι είναι παρόντες και βλέπω ότι ε, έχουμε πολλούς και από τους πρασίνους ε, που είναι στην αίθουσα. Καλά τα έχετε πάει. Αναλογικά τουλάχιστον τα έχετε πάει καλά. Λοιπόν, το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι το 12, βιώσιμη διαχείριση των κοινών με την Νορβηγία και την Ισλανδία θεμάτων. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με το ζήτημα της Ισλανδίας. Θα θυμάστε ότι είχε γίνει μια συζήτηση, αν δεν κάνω λάθο, στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όπου είπαμε ότι η Ισλανδία και η Γρυλανδία μονομερό είχαν αποφασίσει ότι θα είχαν μεγαλύτερο μεγαλύτερη ποσόστοση όσον αφορά το σκουμπρί, στα κοινά αποθέματα πάντα, και φάνηκε τότε ότι και τα αποθέματα για το είδος αυτό, για το σκουμπρί, παρουσίαζαν μείωση, τουλάχιστον υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητά του και είχαμε πει τότε ότι ενδεχομένω θα έπρεπε να ληφθεί κάποια δράση κατά τη Ισλανδία, προκειμένου να έχουμε μια πιο σταθερή και ισότιμη σχέση μεταξύ των συμβαλωμένων μερών και ενδεχομένω θα έπρεπε να ληφθούν και κάποιε κυρώσει κατά τη Ισλανδία. Έκτοτε μάθαμε ότι τα αποθέματα για το σκουμπρί ήταν καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, αλλά αυτό δεν διευθετεί το ζήτημα της ποσόστοσης, όπου φαίνεται ότι η Ισλανδία και η Γρυλανδία επιθυμούν να έχουν μια υψηλότερη ποσόστοση, που αντιστοιχεί τελικά σε υψηλότερο ποσοστό των ε, συνολικών επιτρεπόμενων αλλιευμάτων. Συνεπώς, έχουμε τον Όρμαν Γκρέχαμ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για το ζήτημα αυτό. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας ε, παρουσιάσω κάποιες πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τα κοινά αυτά αποθέματα και τη συμφωνία που έχουμε για το Σκουρμπρί με την Νορβηγία και την Ισλανδία και θα ήθελα να αναφερθώ επίσης και στις διαπραγματεύσεις που είχαμε μεταξύ Νορβηγίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσφατα. Λοιπόν, όντω, α ξεκινήσουμε από τη Ισλανδία και ακούμε έπειτα να μα πείτε για την Νορβηγία. Λοιπόν, θα γνωρίζετε ότι τα αποθέματα για το σκουμπρί την χάνουν ε, αλληλευτική εκμετάλλευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νορβηγία, τι Φερόε νήσου, τη Γρυλανδία και τη Ρωσία. Πρόκειται λοιπόν για ένα αλληλευτικό απόθεμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό από οικονομικής πλευράς για τα ευρωπαϊκά αλληλευτικά σκάφη και αυτές οι παράκτιες χώρες έχουν προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για το απόθεμα αυτό. Στι πραγματεύσει αυτέ όλα τα συμβαλώμενα μέρη συμμετέχουν προκειμένου να συζητήσουν το καθεστώ, την κατάσταση του αποθέματο αυτού και τι μπορεί να γίνει για την καλύτερη διατήρησή του. Δυστυχώς τρία μόνο συμβαλόμενα μέρη, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία και η Φερόε Νήσι έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία διότι η Νορβηγία και η Ρωσία δεν έχουν συνάψει μια συμφωνία όσον αφορά τα κοινά αποθέματα. Από το 2014 υπάρχει αυτή η συμφωνία για τα κοινά αποθέματα που τίθεται ένα ποσοστό 16% για το απόθεμα του Σκουμπρούι το οποίο μπορούν μεταξύ τους να μοιραστούν τα τρία συμβαλώμενα μέρη. Δυστυχώ όμω, οι δραστηριότητε τη Ρωσία, τη Γρυλανδία και τη Ισλανδία υπερβαίνουν αυτό το 16,5% με αποτέλεσμα τελικά τα αλλιεύματα να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Το 2020 παρόλα αυτά περιμένουμε ότι το απόθεμα αυτό θα ανασυσταθεί. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο θεωρούμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Είχαμε λάβει συγκεκριμένες τιμωρητικές κυρώσεις το 2019 αλλά και το 2018 και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί πολύ σημαντικά το συνολικό επιτρεπόμενο αλλιεύμα για το σκουμπρί και εμείς τότε Απευθυνθήκαμε επίσης και στις Φερόες νήσους, ζητώντα τους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Η ΆΙΣΙΣ τον Μάρτιο προχώρησε σε μια συγκεκριμένη επιστημονική πραγματογνωσύνη και έδειξε τελικά η πραγματογνωσύνη αυτή ότι το απόθεμα σκουμπριού ήταν πολύ πιο υγιές από ό,τι είχαμε νωρίτερα εκτιμήσει. Παρ' όλα αυτά, όταν οι παράκτιες αυτές χώρες συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν περαιτέρω τα περί των κοινών αποθεμάτων αποφάσισαν να μην τροποποιήσουν το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα, το τάκ και το σκουμπρί, ότι θα δικαιολογεί το κάτι τέτοιο. Επομένως, αυτή τη στιγμή το τάκ το οποίο έχουμε θα έπρεπε να συνάδει περισσότερο με τη σύσταση της ISIS. Δυστυχώ, όμως, όπως είπατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε, η Ισλανδία προχώρησε σε μια μονομερή απόφαση, όχι μόνο να αυξήσει την ποσόστοσή τη, παραβαίνοντα κατά αυτόν τον τρόπο τα όσα λέει η ISIS, αλλά αποφάσισε να υπερβεί μάλιστα και το ιστορικό απόθεμα, το, μάλλον το, το ιστορικό επιτρεπόμενο αλίευμα, το οποίο προβλέπεται για το σκουμπρί και καταλαβαίνετε ότι αυτό αντιβαίνει στις προσπάθειες που έχουν καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Φερόες Νήσι και η Νορβηγία προκειμένου να καταστήσουν το απόθεμα αυτό βιώσιμο. Είπαμε επίσης ότι η Ισλανδία δεν ε, έχει κάνει κάποιες ε, επίσημες ε, προσπάθειες για να συμμορφωθεί τελικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένουμε ακόμα να λάβει κάποια δράση. Μολονότι λοιπόν δεν συμφωνούμε μετά όσα έχει κάνει αυτή τη στιγμή η Ισλανδία αλλά και η Ρωσική Ομοσπονδία. Οι χώρε αυτέ είναι σε θέση να αιτιολογήσουν τουλάχιστον την στάση του. Αλλά θεωρούμε ότι και πάλι η υπέρβαση του επιτρεπόμενου αλλιεύματο κορμπιού από την Ισλανδία δεν μπορεί να αιτιολογηθεί δεόντω. Υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσα να σα δώσω αυτή τη στιγμή. Πάντω, σήμερα το πρωί υποβάλαμε μία πρόταση προς την συνεδρίαση της Επιτροπής του Βορειοατλαντικού Ωκεανού λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή η συνεδρία αυτή, προκειμένου να τεθεί ένα ανώτατο όριο ως προς αφορά, όσον αφορά την αλίευση του είδους αυτού και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιοριστεί η υπεραλίευση της Ισλανδίας. Γιατί βλέποντας την κατανομή των ποσοστώσεων, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η Ισλανδία αυτή τη στιγμή δεν υπεραλλιεύει μόνο στα δικά της ύδατα, τα Ισλανδικά, αλλά προβαίνει και σε υπεραλλίευση για το σκουμπρί στα διεθνή ύδατα, όπου επιτρέπεται να λιεύει. Επομένως, με, την, με το νέο αυτό όριο το οποίο προτείνουμε σε τόνους, και το οποίο αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται η Επιτροπή του Βορειοατλαντικού, Βορειοανατολικού, με Ατλαντικού, πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε τελικά να περιορίσουμε την αλληλευτική αυτή δραστηριότητα της Ισλανδίας. Πάντως, προφανώς αποδοκιμάζουμε τις δράσεις αυτές της Ισλανδίας και αυτό το θίξαμε δεόντως στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις που είχαμε μαζί τους. Τίθεται το ζήτημα βέβαια της βιωσιμότητας του είδους αυτού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι όλα τα συμβαλώμενα μέρη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις συμφωνηθήσεις ποσοστώσεις. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά το ζήτημα αυτό για το σκουμπρί. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα με αυτά που μας προτείνετε, ακούγοντας ιδιαίτερα αυτά που προτείνετε για τα τάξη τα επιτρεπόμενα όρια λήψης. Αυτά που λέτε είναι πολύ σαφή και πιστεύω ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε όσον αφορά αυτά που συμβαίνουν και στα διεθνή ύδατα αλλά και στα εθνικά τους ύδατα. Και θυμάμαι όταν είχαμε τον Επίτροπο εδώ και έδωσε απαντήσεις, δεν πήραμε απαντήσεις για την Ισλανδία ικανοποιητικές. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν, προσπαθήσατε να έχετε κάποιες απαντήσεις είχατε κάποια ανταπόκριση. Εμάς πάντως οι απόπειρέ μας να έχουμε μαζί τους συνεννόηση να έρθουν εδώ στην Επιτροπή δεν καρποφόρησαν. Όλες μας οι προσπάθειες ε, δεν είχαν ε, αποτέλεσμα. Εσείς μπορείτε να μας δώσετε μία παρουσίαση του τι προσπαθήσατε, τι κάνατε και τι αποτέλεσμα είχατε. Επίσης κατάλαβα ότι κάνατε μια πρόταση στην Επιτροπή του Βόρειο Ατλαντικού, αλλά πώς μπορούμε να επηρεάσουμε το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την ερώτηση που κάνετε. Τώρα, πόσες φορές πλησιάσαμε την Ισλανδία. Ναι, έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές από τότε που ξεκίνησε, από το 18-19. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, ιδιαίτερα ε, όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα ήδη από το 11-12 με την υπεραλίευση. Και είχαμε πολλές επαφές τεχνικού επίπεδου, δύο φορές το χρόνο και σε ψηλότερο επίπεδο, υπουργικό ε, επίπεδο, όπου εμείς από την Επιτροπή θελήσαμε να τους κάνουμε κάποιες προτάσεις και περιμέναμε τις αντιπροτάσεις τους. Πρέπει να σας πω ότι πάντα η Ισλανδία απαντούσε ναι, θέλουμε να συμμετέχουμε, αλλά συγκεκριμένη πρόταση ή αντιπρόταση δεν λάβαμε ποτέ. Και είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία έχουν αναπτύξει ήδη από τη δεκαετία του 70 κάποιες κοινέ δραστηριότητες και η Ισλανδία ποτέ δεν συμμετείχε. Πρέπει να σας πω ότι οι σχέσεις μας με την Νορβηγία είναι εξαιρετικά σημαντικοί και νομίζω ότι λειτουργούμε με κάποια κοινά αποδεκτά πρότυπα. Αλλά από τη μεριά της Ισλανδίας δεν είχαμε ποτέ ανταπόκριση και το Σεπτέμβριο όταν ξεκίνησαν οι νέες διαβουλεύσεις ε, η Ισλανδία είπε ναι θέλουμε να συμμετέχουμε κι εμείς αλλά επαναλαμβάνω δεν είχαμε συγκεκριμένα στοιχεία. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά δύσκολο να σας πω ότι κάτι απτό έχει προκύψει από όλες αυτές τις συζητήσεις και τον ε, διάλογο. Τώρα, όσον αφορά την Επιτροπή του Βόρειο Ατλαντικού, περιμένουμε να δούμε τα άλλα μέρη και τα άλλα, τους, οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, η Ρωσία, η Γρυλανδία, η Ρωσία, από αυτούς, αν θέλετε, εξαρτάται και από τη δυναμική που θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε. Αν έχουμε πλειοψηφία που υποστηρίζει την πρότασή μας, σαφώς και θα προχωρήσει η πρότασή μας. Αλλά επειδή είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός, πρέπει να περιμένουμε τους υπόλοιπους για να δούμε τι κατεύθυνση θα πάρει αυτή η συζήτηση. Υπάρχει θέμα συζήτησης ε, για κυρώσεις κατά της Ισλανδίας. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για κυρώσεις, <clears throat> γιατί υπάρχουν κάποια, αν θέλετε, εμπόδια τα οποία θα πρέπει να ξεπεράσουμε για να δείξουμε ότι δεν είναι βιώσιμη αυτή η αντιμετώπιση, ότι δεν υπάρχει συνεργασία, δεν υπάρχει απροθυμία Μέχρι τώρα πρέπει να σας πω ότι οι προσπάθειές μας όντως έχουν αντιμετωπιστεί με θετικό τρόπο μεν, αλλά χωρίς τίποτα το συγκεκριμένο και το απτό. Και βεβαίως όσον αφορά την βιώσιμη αλληλεία βεβαίως και αυτή η δραστηριοποίηση και η υπεραλλίευση από μέρους της Ισλανδίας είναι πάρα πολύ αρνητικά και λυπηρά φαινόμενα πρέπει να μας ε, υποβάλουν, μάλλον να υποβάλουν στην Επιτροπή του Βορείου Ατλαντικού τα μέτρα που έχουν λάβει για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων. Είναι δύσκολο πάντως να μιλήσουμε για κυρώσεις. Θα πρέπει να έχουμε και την προσέγγιση μέσω της Επιτροπής του Ατλαντικού. Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε και εκεί τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι κάνετε ό,τι μπορείτε, το φαντάζομαι. Αλλά οι Ευρωπαίοι αλληλείς θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι ε, δεν θα χρειαστεί να ξανάρθετε εδώ πέρα στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσετε κάποιο εναλλακτικό σχέδιο, αλλά ενδεχομένως με το νέο έτος να χρειαστεί να κάνετε κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά την Νορβηγία, Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ πέρα να καλύψουμε και τη χώρα αυτή, γιατί η κυρία Κέρσεν που κάθεται δίπλα σας μας είπε πριν από λίγο καιρό ότι έχουμε 81, 81 αποθέματα τα οποία παρακολουθούμε, 59 αποτελούν αντικείμενο κοινών αποθεμάτων με την Νορβηγία. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιπαράθεση με τη χώρα αυτή και τι κάνουμε για να επιληθούν τα κακό κείμενα. Πιστεύω ότι είναι καλό να δούμε και αυτό το θέμα σε σχέση με την ε, ε, Νορβηγία. Βεβαίως δεν υπάρχει ε, συμφωνία για πολλά από τα πελαγικά ή βανθυπελαγικά είδη, αλλά αυτό δεν έγινε επειδή εμείς δεν έχουμε κάνει προσπάθειες. Ελπίζουμε ότι θα στεφθούν από επιτυχία οι οποίες προσπάθειες έχουμε κάνει μέχρι του χρόνου οι διαβουλεύσεις ε, με την ε, Νορβηγία αφορά ε, την, περιοχή Σκάγκερακ και την Βόρεια Θάλασσα και βεβαίως αφορά τα πεθυπελαγικά είδη όπως είναι ας πούμε η χωματίδα, όπως είναι το σκουμπρί. Η διαδικασία που θα ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα ήδη από την Δευτέρα θα είναι να μελετήσουμε καλύτερα τις ε, ε απόψεις και τις προτάσεις ε, των επιστημόνων, να δούμε τι έχει να μας πει η νορβηγική πλευρά και ενδεχομένως να υποβάλουμε τον Δεκέμβριο εμείς ε, μαζί με το Συμβούλιο μια πρόταση. Ιστορικά είχαμε ε, διαχείριση των αποθεμάτων βάσει της λεγόμενης μακροχρόνιας διαχείρισης αποθεμάτων. Με τα χρόνια όμως ε, αυτό ε, έγινε στην ουσία φάνηκε ότι είναι λίγο απορχαιωμένο γιατί άλλαξαν οι επιστημονικές απόψεις, άλλαξαν και τα πολιετή σχέδια διαχείρισης και επομένως θα έπρεπε αυτό το, αυτές οι στρατηγικές μακροχρόνιας διαχείρισης να αναθεωρηθούν. Και άλλωστε μην ξεχνάτε ότι στόχος μας ε, είναι ε, να έχουμε όσο γίνεται πιο σύγχρονες και επικαιροποιημένες συμφωνίες. Ιστορικά λοιπόν όντως κάποια από τα αποθέματα ε, αλλιεύονται βάση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Θα δούμε όμως πώς έχουν εξελιχθεί οι καταστάσεις και αυτά θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα στις συζητήσεις. Έχουμε μια κατάσταση που σε γενικό επίπεδο λέμε ότι σε γενικές ε, λέμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη γνώμη των, επιστημόνων καθότι έχουμε σταδιακή μείωση κάθε χρόνο όμως σταθερή σταδιακή ε, ε μείωση ε, ας πούμε ε, και για το σκουμπρί καθώς επίσης και για τον be heading towards a situation where all the jointly managed stocks in Norway will be will be set at FMSY. But I would like to note καθώς επίσης και για κάποια άλλα είδη δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου όσον αφορά τις συμφωνίες μας. Ξέρω όσον αφορά όμως τα άλλα ε, όπως ας πούμε για τον νορβηγικό βακαλάο, Norway Pout, ε, μαζί με την FMSY ε, η κατάσταση εδώ είναι λίγο διαφορετική. Έχουμε αυτές τις συμφωνίες, δεν είναι όπως με τον Γελφίνο. Όσον αφορά τώρα τον Γάδο, είναι η κατάσταση η οποία πιο πολύ μας προβληματίζει. Θέλουμε να ακολουθήσουμε την επιστημονική ε, πρόταση ε, για μείον 61% ε, αλλιευτική ικανότητα για την επόμενη χρονιά. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και για τον Εγγελφίνο είναι σημαντική, σημαντικό ποσοστό. Στόχος μας είναι είναι να ε, υποβάλουμε επιπλέον ε, μέτρα, μια και αυτή είναι άλλωστε η υποχρέωσή μας. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τους επόμενους μήνες ποια είναι τα μέτρα, τα συνοδευτικά, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθούν έτσι ώστε να προκύψει ανασύσταση του αποθέματος γάδου. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και κάποιες τεχνικές, ε, ε, κάποιους τεχνικούς ε, κανονισμούς για τα νορβηγικά ύδατα και τα ευρωπαϊκά ύδατα, έτσι ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες level playing field για όλα τα σκάφη τα οποία αλλιεύουν στην περιοχή. Είναι σημαντικό όσο γίνεται πιο γρήγορα να εισαχθούν τα μέτρα αυτά και θα, θα θέλαμε πραγματικά αυτό να γίνει μέσω κατεξουσιοδότηση πράξης. θα, θα δούμε βεβαίως και ε, τι απόφαση θα πάρει και το Κοινοβούλιο. Εν συνόψη, εμείς ε, ε, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπλέον πιέσεις και επομένως να πάρουμε τα απαραίτητα συνοδευτικά μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος από τα μέλη να πάρει το λόγο. Όχι. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, λέει ο Πρόεδρος, ε, θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τα μέγιστα επιτροπόμενα αλλιεύματα, αλλά για τα περισσότερα από θέματα μάλλον θα μπορέσετε ε, να ε, υποβάλλετε κοινέ προτάσεις. Ναι, την επόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες διαπραγματεύσεις και τον Δεκέμβριο θα αρχίσουμε να ξεκινήσουμε την επεξεργασία πρότασης. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Αυτά είναι όλα πάρα πολύ θετικά πράγματα και επομένως συνεχίζουμε. Προχωράμε, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Είχα πει στην αρχή της χθε, χτεσινής συνεδρίας ότι θα αλλάξουμε λίγο την ε, σειρά και επομένως ε, επόμενο θέμα ε, θα είναι η ετήσια οικονομική έκθεση ε, για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Στόλου. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ. Σας ευχαριστώ για την θέση σας. Σας καλωσορίζουμε σε αυτήν την επιτροπή μας η οποία έχει λίγο αποδεκατιστεί φοβούμε. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ πολύ. Ε, ούτως ή άλλως ε, το ε, δεν είναι θέμα ποσότητας, είναι θέμα ποιότητας και εδώ είμαστε λίγοι αλλά καλοί. Λέει ο πρόεδρο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε έτσι ώστε να αναφερθώ στο θέμα αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον νομίζω γιατί αναφέρεται σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Λοιπόν, εδώ αναφερόμαστε στα οικονομικά της αλληλευτικής πολιτικής στην ουσία και θα ήθελα ε, να πω το εξής. Μιλάμε διαρκώς για βιωσιμότητα ε, απέναντι ή σε αντιδιαστολή μάλλον με την οικονομική εμπορική δραστηριότητα, ενώ στην ουσία μιλάμε για ένα και το αυτό. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ε, ότι και τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά εξαρτώνται από την ε, βιωσιμότητα και ελπίζω να μπορέσω εδώ να σας ε, καταδείξω αυτήν την σχέση. Περί ε, συζητούμε. Μιλάμε στην ουσία ε, για την ε, έκθεση που έχει το όνομα έκθεση ε, για τον αλλιευτικό στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως γίνονται τελείως διαφορετικές εκθέσεις για τα επιμέρους τμήματα. Ξέρετε ότι υπάρχει και ένα μακροοικονομικό παρατηρητήριο που παρακολουθεί τις τιμές, τις τιμές αγοράς ε, και πώλησης. Εδώ βλέπετε μία συνολική εικόνα. Ο μιλητής λέει ότι προβληματίζομαι λίγο γιατί δεν είναι ακριβώς αυτή η παρουσίαση που θα ήθελα να κάνω. Δεν πειράζει. Αφού σας έδειξε τη διαφάνεια αυτή να το συνεχίσω, βλέπετε εδώ λίγο μια γενική εικόνα του πώς έχουν τα πράγματα. looks Ωραία. Τώρα έχουμε τις σωστές διαφάνειες. Πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς χωρίζουμε τον ε, στόλο σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Βλέπετε εδώ στη διαφάνεια ε, υπάρχει μια, ε, μια σχετική ισορροπία όσον αφορά τους, ε, τις ε, θέσεις εργασίας, αλλά μετά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Εάν δείτε τώρα την κατάσταση ανά χώρα όσον αφορά τις θέσεις εργασίας στον ελευτικό τομέα, ε, βλέπουμε βέβαια τις μεγάλες χώρες της ε, Μεσογείου, ε, από την άλλη μεριά ε, στην Ελλάδα ας πούμε υπάρχουν μονάχα 30.000 σκάφη με 15% όμως αντιπροσώπευση όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Ποια είναι τώρα η συνολική εικόνα. Η έχει βελτιωθεί και ε, η αποδοτικότητα, η κερδοφορία δηλαδή και ε, οι απολαβές από την δραστηριότητα. Εμείς κάνουμε αυτή την οικονομική ε, έρευνα εδώ και πολλά χρόνια και είμαστε σε θέση επομένως να δούμε τάσεις και να ερευνήσουμε τις τάσεις ε, αυτές. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μία συνεχής ε, περίοδος σημαντικής ανάπτυξης. Αλλά βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος που όλα δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Εξακολουθούμε να έχουμε απώλειες όσον αφορά τον ευρωπαϊκό στόλο και υπάρχουν τέσσερις εθνικοί στόλοι οι οποίοι έχουν υποστεί ιδιαίτερες απώλειες ε, την τελευταία χρονιά. Βλέπετε εδώ ποιες είναι αυτές οι τέσσερις χώρες. Ε, βέβαια δεν είναι θέμα συγκυρίας. Ε, πρόκειται για στόλους οι οποίοι δρούν σε περιφέρειες με μείωση της βιωσιμότητας. Αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι της διασύνδεσης που θέλω να κάνω ανάμεσα στην ελευτική διαδικασία και τη βιωσιμότητα. Η Μεσόγειος επίσης έχει μείνει πάρα πολύ πίσω όσον αφορά ε, σε όρους δηλαδή οικονομικής ε, αποδοτικότητας ε, και Έχουμε εδώ μία σαφή μειωτική τάση που μπορεί να είναι βεβαίως το, ο να έχει πολλά στοιχεία που οδηγούν σε αυτήν, βιομηχανική δραστηριότητα, γενικότερη κατάσταση αποθεμάτων κλπ. Όσον αφορά το μέλλον πάλι, εδώ ε, πραγματικά υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο διαρκώς βαίνει βελτιούμενο όσον αφορά ε, την ε, βιωσιμότητα και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε όλα τα μέτρα συντήρησης. Εδώ βλέπετε κυρίως ε, θέματα τα οποία αφορούν ε, την Βόρεια Θάλασσα και τον ε, Ατλαντικό και σε όρους όγκου 98% της 100 των αλλιευμάτων 98, 98 α αναφέρεστε στον όγκο των εκφορτωμένων ψαριών. Um, ε, έλεγα προηγουμένως ότι η μεγάλη εικόνα είναι θετική. Βλέπουμε ότι ε, ο αλλιευτικός στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι αποδοτικός, έχει ένα περιθώριο μεικτό περιθώριο κέρδους για το 17-25,8% ε, και το καθαρό ε, περιθώριο για το 17 ήταν 1,34 δις, ε, δηλαδή πέντε φορές παραπάνω από το αντίστοιχο ποσό του 2008. Δεύτερο στοιχείο, ο κλάδος της αλίας κάνει σημαντικές επενδύσεις. Επενδύει λοιπόν ο κλάδος στην περίοδο 2008-2017 είχαμε 8,31 δις ευρώ που επενδύθηκαν το 17 δε 551 ε, εκατομμύρια. 3 ε, ε, δις αναφέρονται μονάχα στα σκάφη, στις αδειοδοτήσεις κλπ. Μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια και για το Ταμείο Διαχείρισης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαχείρισης της ε, Αλίας, που βεβαίως συμβάλλει σε αυτές τις επενδύσεις. Είχαμε ε, σημαντική αύξηση και της παραγωγικότητας ε, και των απολαβών και των μισθών αλλά όπως είπα και ε, προηγουμένως, ενώ ε, αυξάνεται, αυξάνονται ε, οι μισθοί, έχουμε μείωση όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Ενδεχομένως θα είναι από τους κλάδους που στο μέλλον δεν θα δούμε πολύ μεγάλες αυξήσεις όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γιατί για να δημιουργηθούν θέσει εργασία χρειάζονται ε, πολλαπλά στοιχεία τα οποία εδώ φαίνεται ότι δεν τα έχουμε. Ε, μικρής κλίμακας ε, αλία, αυτά τα σκάφη πάνε καλύτερα, αυτός ο κλάδος δηλαδή έχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά μένει ακόμα πίσω κυρίως όσον αφορά το εντατικό βιομηχανοποιημένο κομμάτι της αλλιευτικής ε, δραστηριότητας. Επίσης η μισθή εδώ είναι χαμηλότερη από το μέσο 17.000 ε, αναέτος μέσο όρο έναντι 28.000. Και βεβαίως αναπτύσσεται και με πιο αργό ρυθμό. Δεν θέλω να σταματήσω ακριβώς, αλλά πρέπει να σας ε, ευχαριστήσω ε, δεν μπορούσα να αναφερθώ σε όλο το έγγραφο. Είναι πάρα πολλών σελίδων το έγγραφο αυτό. Έχουμε μια ολόκληρη ομάδα η οποία ασχολείται με, τα, ε, με τη σύνθεση αυτή. Μιλάμε για ένα τομέα για τον οποίο έχουμε πάρα πολλά ε, δεδομένα. Πρέπει να σας πω ότι πριν από τρεις εβδομάδες αναγκαστήκαμε να πάρουμε και πολύ δύσκολες αποφάσεις στο Συμβούλιο αλίας. Ε, πρέπει να δούμε τα στοιχεία, πρέπει να κάνουμε οικονομική ανάλυση, πρέπει να καταλάβουμε, να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα οποία αποφασίζουμε, τα μέτρα που παίρνουμε είναι αποδεκτά και βάση της επιστήμης αλλά και βάσει των οικονομικών αναγκών ε, και απαιτήσεων του κλάδου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας λέω αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε ενδεχομένως να μελετήσετε κάποια εξειδικευμένα τμήματα, κάποιες εξειδικευμένες περιοχές, παρακαλώ μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή με μένα. Μια ερώτηση να κάνω. Αυτή η κερδοφορία τελικά είναι θετικά νέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που είναι τόσο χαμηλές οι τιμές των καυσίμων και που ουσιαστικά αυτό δεν συνάδει τόσο πολύ και με τους στόχους που έχουμε θέσει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Δεν σχετίζεται άμεση η αύξηση των τιμών με τη μείωση της κερδοφορίας και το αντίστροφο. Έχετε απόλυτο δίκιο, όντως, ένας βασικός παράγοντας του κόστους είναι οι τιμές των καυσίμων. Αυτό επηρεάζει το σύνολο του κλάδου, αναμφίβολα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όταν μειώνονται οι τιμέ των καυσίμων, αυξάνονται τα κέρδη και το αντίστροφο. Το άλλο ζήτημα βέβαια που τίθεται είναι πώ να εξηγήσουμε τι μακροχρόνιε τάσει. Στον πίνακα αυτό που σα έδειξα, αν έβαζα μια καμπύλη για την τιμή των καυσίμων, θα βλέπετε μια συνεχή διακύμανση, μια συνεχή πτυτικότητα των τιμών αυτών, που σαφώ επηρεάζει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά όχι με τρόπο καθοριστικό. Και βέβαια, ξέρετε ότι η βιώσιμη αλία σε βάθος χρόνου είναι πολύ πιο επικερδής, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν αλλιεύει κανείς με έναν τρόπο πιο βιώσιμο, τελικά καταφέρνει να εξοικονομήσει και σε τιμές καυσίμων αλλά και σε κόστος εργασίας. Βλέπετε λοιπόν ότι ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει πάρα πολύ την κερδοφορία σε βάθος χρόνου είναι η βιωσιμότητα της εταιρεία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ήθελα καταρχήν να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την τόσο θετική παρουσίαση. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε λάβει υπόψη και τις μελλοντικέ προοπτικές όσον αφορά τη Βόρεια Θάλασσα. Εγώ είμαι από την Ολλανδία και στην Ολλανδία και στη Γερμανία έχουμε ανεμογεννήτριες και έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική βιοπικιλότητα στα πλαίσια του Natura 2000. Και αυτό ισχύει για πολλές χώρες Ευρώπης. Μπορούμε να κρατήσουμε αυτές τις θετικές πτυχές που μας παρουσιάσατε παρόλα αυτά. Όσον αφορά τώρα την ε, ερασιτεχνική αλία, την ε, αλία η οποία δεν είναι επαγγελματική, μπορούμε να τηρήσουμε τους στόχους αυτούς όπως προβλέπονται από την κοινή αλληλευτική πολιτική, γιατί και αυτός ο τομέας είναι σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πρέπει να δούμε την πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Εγώ εκπροσωπώ εδώ το τμήμα αυτό της Επιτροπής Αλίας και αν κοιτάξω γενικότερα το θαλάσσιο περιβάλλον υπάρχουν πολλές διαφορετικές, αν θέλετε, ανταγωνιστικές θάσεις ε, και ο τομέας της απασχόλησης 150.000 θέσεις απασχόλησης ε, στον τομέα της αλίας ο αριθμός αυτός ε, μειώνεται και αντίθετα βλέπουμε τον τομέα της ε, πολύ συγκεκριμένη ηχθειοκαλλιέργεια, παραδείγματο χάρη, 210.000 ε, νέε θέσει απασχόληση δημιουργήθηκαν και σε παρεμφερή επαγγέλματα. Βλέπετε λοιπόν ότι σε πολλούς τομείς υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν νέε θέσει απασχόλησης όσον αφορά την αεραστεχνική αλία, την αλία ψυχαγωγία. Και στην Δανία και στη Σουηδία και στις κάτω χώρες και στη Γερμανία. Σίγουρα υπάρχει εδώ περισσότερη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα της αεραστεχνικής αλίας και τι θέλουμε να κάνουμε για να παραμείνει ζωντανός αυτός ο τομέας. Όλα αυτά που αφορούν την αεραστεχνική αλληλεία, ενοικίαση σκαφών, το τουριστικό κομμάτι, τα ξενοδοχεία, η εστίαση, όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, γιατί όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά και δραστήρια. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω δύο σημεία. Μιλήσατε για τις τιμές των προϊόντων, κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για έναν υγιή και δυναμικό τομέα. Πολλές φορές όμως δεν δίνουμε αρκετή συμμαχία στην τιμή πώλησης των προϊόντων αυτών και γιατί ξαφνικά αυξάνεται η τιμή τους. Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι εξηγήσει οι αιτιολογίες λείπουν και στην παρουσίασή σας μάλιστα θα θέλαμε να έχουμε λίγο μία λίγο πιο λεπτομερή παρουσίαση όλων αυτών των στοιχείων που αφορούν την τιμή, τη διάθεση στην αγορά, την πρόθεση αυτών των προϊόντων. Από τη στιγμή δηλαδή που θα γίνει η εκφόρτωση μέχρι τη στιγμή που θα διοχετευτεί στην αγορά το συγκεκριμένο προϊόν. Συντήρηση, μιλήσατε για κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε και θα προτιμούσα να μου λέγατε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, ότι οι πολιτικές διατήρησης που έχουν υιοθετηθεί δεν συμβάλλουν στα αρνητικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν αυτό που λέτε πάντως ε, στηρίζεται σε πραγματικές ε, αποδείξεις ή αν είναι μια απλή δήλωση. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, ευχαριστώ πολύ και αν θέλετε θα σας φέρω σε επαφή με κάποιους από τους συναδέλφους οι οποίοι είναι ίσως πιο αρμόδιοι από μένα και θα σας δώσουν στοιχεία για το κομμάτι της διάθεσης στην αγορά, το marketing και σίγουρα η αύξηση των τιμών είναι κάτι που τους απασχολεί και που το έχουν επεξεργαστεί. Τώρα, τι στοιχεία έχουμε που να στηρίζουν την άποψη ότι η βιώσιμη αλληλεία δεν έχει μόνο αρνητικές αλλά και πολλές θετικές ε, επιπτώσεις. Έχουμε εργαστεί, έχουμε κάνει ανάλυση οικονομετρική, ανάλυση στοιχείων και πολλοί συνάδελφοι έχουν επεξεργαστεί βάθος το θέμα αυτό μία δεκαετία νομίζω μας απασχολεί το θέμα αυτό και έχουμε στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να δηλώσουμε με ακρίβεια ότι υπάρχουν και θετικές συνέπειες. Αν θέλετε, αυτό είναι η περίληψη, λέει ο πρόεδρος του συνολικού εγγράφου. Έχουμε και το σύνολο των στοιχείων. Και για τη Μεσόγειο, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι ο στόλος που δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βελτιώνει το 2017 με αυξημένα κέρδη, με διακυμάνσεις βέβαια μεταξύ των ε, χωρών. Ο πιο σημαντικός τόλος είναι ο Ιταλικός, ο οποίος και παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την αύξηση των κερδών και μιλάμε και για τις αυξημένες εκφορτώσεις. Μα εγώ νομίζω ότι υπήρχε υπεραλίευση Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο περίπλοκη η κατάσταση και ότι η αύξηση των εκφορτώσεων Μα θα πρέπει κάθε φορά να δούμε για ποια περιοχή μιλάμε, για ποιο αλλιευτικό απόθεμα. Ο Ιταλικός στόλος, ναι, σίγουρα παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Μεσογείου. Επιτρέψτε μου όμως να κοιτάξω πολύ συγκεκριμένα τα στοιχεία αυτά και να σας δώσω μια απάντηση που να βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία, σε αριθμούς. Ευχαριστώ. Α, συγγνώμη κύριε Παντέλα, δεν σας είχα Ευχαριστώ πρόεδρε. και σας ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Από την παρουσίαση αυτή είναι σαφές ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο και με την αλία μικρής κλίμακας, την παραδοσιακή αλία, γιατί είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τα ποσοστά αλίευσης τα οποία αναλύουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι σαφές ότι θα πρέπει και ο κλάδος αυτός πέρα από τη βιομηχανική δηλαδή να μας απασχολήσει. Εγώ είδα την πολυσέλιδη αυτή έκθεση και το πιο ενδιαφέρον θεωρώ είναι ότι γίνεται μια αναφορά και στις κάτω χώρες. Στην έκθεση πάντως αυτήν, δεδομένου των υποχρεώσεων εκφόρτωσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, συγκεκριμένα είδη τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αναφέρουμε στο καλκάνι για παράδειγμα. Γίνεται μία αναφορά στην έκθεση στο είδος αυτό και λέτε ότι ε, μπορούμε να περιμένουμε ότι μέσω των ειδών αυτών θα επηρεαστούν πολύ αρνητικά κάποιοι αλλιευτικοί στόλοι που ορισμένοι θα καταφέρουν να καν αλλιεύουν πλέον. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και στα ίδια αυτά. Κάθε φορά λοιπόν που πρέπει να συμμορφωθούμε με τι υποχρεώσει που προβλέπονται για αυτά τα είδη, όπω το καλκάνι, α μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι αλληλευτικοί στόλοι που επηρεάζονται πολύ αρνητικά και οι δεν μπορούν να βγουν καν στα ανοιχτά. Αυτό δεν αφορά μόνο τι κάτω χώρε, αλλά κυρίω τι κάτω χώρε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η ακόλουθη. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αποφύγουμε τα ίδια αυτά τα οποία αναφέρεται όπως το καλκάνι να φέρουν σε τόσο δύσκολη θέση συγκεκριμένους αλληλευτικούς στόλους. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ πολύ να μας διαφωτίσετε ως προς αυτό πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια τόσο αρνητική κατάσταση για κάποιους ελευτικούς στόλους. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ως αριθμιστικές αρχές, αλλά και ως απλοί πολίτες, θα πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιό μας περιβάλλον με κάθε δυνατό τρόπο, με έναν τρόπο πολυδιάστατο. Και βέβαια αναφέρομαι και στα ίδια εκείνα, τα οποία βρίσκονται σε πολύ δεινή κατάσταση. Και ξέρετε ότι το έργο αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι ε, σαφώς μέσω των μέτρων αυτών συντήρησης επηρεάζονται συγκεκριμένοι ελευτικοί στόλοι. Και πολλές φορές ε, ξέρετε ότι ε, αλλιεύουμε ένα συγκεκριμένο είδος, αλλά στα δίκτυα μας πιάνουμε και πολλά άλλα είδη, τα οποία δεν στοχεύαμε, τα οποία δεν θα έπρεπε να λιεύουμε, διότι κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Αναφερθήκατε σε κάποια είδη γάδου, αναφερθήκατε επίσης στο καλκάνι, είδη τα οποία παρουσίασαν πολύ αρνητικά αριθμητικά δεδομένα φέτος. Αναφερόμαστε εδώ πέρα βέβαια σε καταστάσεις που μας υποχρεώνουν να υποβάλουμε συγκεκριμένους περιορισμούς όσον αφορά τις αλληλευτικές δυνατότητες. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι σαφώς δεν είναι εύκολο να πάρει κανείς τέτοιες δύσκολες αποφάσεις όταν εν γέννη ο λευτικός στόλος τα πηγαίνει καλά. Γνωρίζετε όμως για ποιους λόγους έπρεπε να ληφθούν τα μέτρα αυτά και κάθε φορά που το Συμβούλιο λαμβάνει τέτοια μέτρα, κάθε φορά που υιοθετούμε τέτοιε αποφάσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώ μπορούμε να μειώσουμε τι ελευτικέ δυνατότητε για τα συγκεκριμένα είδη, αλλά πώ μπορούμε να κάνουμε και την ίδια την αλία πιο επιλεκτική, αποφεύγοντα την παρεπίπτουσα αλία. Είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο μέσω συγκεκριμένων τεχνικών μέτρων και τεχνικών διευθετήσεων και θεωρώ ότι σαφώς έχουμε οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες όμως είναι απόλυτα δικαιολογημένε. Όσον αφορά τον γάδο, όσον αφορά το καλκάνι και τα άλλα είδη στα οποία αναφερθήκατε, σαφώς μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να τροποποιηθεί ο λιευτικός εξοπλισμός, να γίνει η αλληλεία πιο επιλεκτική και να καταφέρουμε τελικά να αποφύγουμε την αλίευση των ειδών αυτών. Και ξέρετε ότι πέρυσι το Συμβούλιο ενέκρινε συγκεκριμένε ποσοστώσει όσον αφορά την αλία για να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην αλλιεύουμε τα ίδια αυτά σε κάθε περίπτωση. Κατά περίπτωση πάντως κάνουμε μία ανάλυση και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ευθύνη μας πάντως είναι να προστατεύσουμε και τα ίδια εκείνα, ιδίως τα ίδια εκείνα, τα οποία από βιολογικής πλευράς αντιμετωπίζουν πολλέ δυσκολίε. Προέδρο. Σαφώ το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο. Α ακούσουμε μία ακόμα ερώτηση. Η κυρία Νταμάτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημείωσα σε αυτά που άκουσα ότι για τη Μεσόγειο ε, η αεραστεχνική ελιοστόλος της ε, αντιπροσωπεύει 72% του στόλου, 51% της ε, απασχόλησης, αλλά μονάχα 22% του αλλιεύματος. Ε, άρα, είναι λογικό να λέω ότι πρέπει να εκπλήσεται κανείς που οι νέες γενιές πλέον δεν θεωρούν ελκυστική αυτή τη δραστηριότητα, άρα, πρέπει, άρα κινδυνεύουμε να χάσουμε μία πολυετή αιωνόβια μπορώ να πω δραστηριότητα η οποία βοηθάει και στην επιλογή 18,4% ε, χρησιμοποιούμε από το Ταμείο Θαλάσσια τους μικρούς ε, Έλλης, όσον αφορά την ε, αλλιευτική προσπάθεια. Βλέπουμε ότι η πίεση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο εξακολουθεί να είναι υψηλή, αλλά βελτιώνεται. Ε, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα όσον αφορά ε, τις αναφορές, αλλά ε, γίνεται λόγος σημαντική μείωση από 12% στο 9%. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε για να, προστατεύουμε την, να προστατέψουμε την ερασιτεχνική αλληλεία. Ολοκληρώνω ερωτώντας το εξής. Εάν λοιπόν από τη μία πλευρά η αλλιευτική ικανότητα έχει μειωθεί ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 1990, αλλά η τάση των ε, τρίτων χωρών της Μεσογείου πάντα, κυρίως οι παρόχθιες, ε, ακολουθούν τελείως διαφορετικό μοντέλο. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή, πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ομοιογενή κατάσταση, κυρίως όταν σε αυτές τις ε, παρόχθιες τρίτες μεσογειακές χώρες έχουμε και κοινωνικό dumping. Uh, Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Εγώ θα έλεγα ότι όσον αφορά τις προκλήσεις και όσον αφορά την ανάγκη να είμαστε πραγματικά προληπτικοί και να προβλέψουμε τι θα γίνει με αυτό το στόλο και συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν πολλές καλές και ελκυστικές θέσεις απασχόλησης, όχι μόνο όσον αφορά το θέμα των εσόδων, αλλά και όσον αφορά την τήρηση των παραδόσεων και των κοινωνικών ιστών. Πρόσφατα υπήρξε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για να υπάρξει και ομοφωνία γύρω από τις ε, χώρες της ε, Μεσογείου αλλά και όσον αφορά το θέμα της ε, ατζέντα για την αλία στη Μεσόγειο. Βεβαίως, για να φτάσουμε σε πραγματικά βιώσιμη αλία, έχουμε πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Είναι μια μακροχρόνια προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν θέλω να σας παρουσιάσω μια καλύτερη, καλύτερη όπως είναι. Και δεν θέλω τώρα να δώσω καλούς και κακούς βαθμούς σε καλούς και κακούς μαθητές. Να μιλήσουμε για τη Βόρεια Θάλασσα, για την Ορβηγία, αλλά κάθε φορά που υπάρχει βιώσιμη αλλήλεια εδώ και πολλά χρόνια, τα πράγματα διαρκώς βελτιώνονται, οι θετικές επιπτώσεις πολλαπλασιάζονται και όντως θα πρέπει να συνεργαστούμε εδώ και με τους εταίρους μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι αυτό είναι το τελικό σας μήνυμα. Υπάρχουν ε, σίγουρα χώρες ε, για τις οποίες στον κλάδο αυτό τα αποτελέσματα δεν είναι πάρα πολύ θετικά. Αλλά η γενικότερη εικόνα είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς την βιώσιμη ανάπτυξη, τα πράγματα είναι καλύτερα. Uh, το επόμενο θέμα είναι το 13, το οποίο έχει αλλάξει αριθμό και είναι το 14. Πρόκειται για τον κυτρινόπτερο τόνο. την υπεραλίευση στον Ινδικό ωκεανό. Είναι ένα είδος το οποίο ήδη έχει υποφέρει από την υπεραλίευση. Το θέμα είναι το πώς αντιμετωπίζονται οι εταίροι μας και το πώς αντιμετωπίζουν κυβερνήσεις όπως αυτή της Νότιας Αφρικής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Θα δώσω το λόγο στην ε, Επιτροπή. Σας καλωσορίζουμε. Θέλετε να μας κάνετε μια πρώτη παρουσίαση. I'm, I'm Ευχαριστώ. Είναι και η τρίτη φορά που παίρνω το λόγο σε αυτήν την Επιτροπή. Πρόκειται για κάτι που αφορά τον έλεγχο, αλλά όχι και μόνο αυτό. Θα σας δώσω καταρχήν λίγα στοιχεία. Περί τίνος πρόκειται. Ο κυτρινόπτερος τόνος είναι ένα από τα τρία είδη του τροπικού τόνου που αλλιεύεται σε διάφορους ωκεανός στην περιοχή και αναφερόμαστε εδώ στον Ινδικό ωκεανό ειδικότερα και πρόκειται για αλεία από αλλιευτικά ε, σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των ποσοστώσεων όσον αφορά τη Γαλλία και την Ισπανία στον Ινδικό ωκεανό είναι το αντικείμενο αυτής της ε, παρουσίασης. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι η αλληλεία του κυτρινόπτερου τόνου ρυθμίζεται από μια διαχείριση IUTC, τοπική διαχείριση αλλιευμάτων, η οποία το 2017 μετά από ένα ψήφισμα που αντικαταστάθηκε από το 18 ένα ψήφισμα του 2018 και τα εμπλεκόμενα μέρη, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν να μειώσουν τις προσπάθειές τους, την αλία τους και την αλίευση στην περιοχή. Το ψήφισμα αυτό όμως δεν ισχύει για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του IUTC, αλλά σε κάποια μόνο, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 21% είναι το ποσοστό που ανήκει που αντιστοιχεί συγγνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά αυτά τα ε, αλλιεύματα. Τα στοιχεία του 2017 ορίζουν ότι το ποσοστό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 50 με 51%. Τώρα, το 15% των ε, ειδών που ελεύονται εκεί είναι ο κυτρινόπτερος τόνος μετά από απόφαση του Συμβουλίου του 2018, η απόφαση 120 ορίζει σε 77.690 τόνους ε, τον κυτρινόπτερο τόνο η ποσόστοση αυτή μοιράζεται κατά 59% στην Ισπανία, στη Γαλλία 39% και το υπόλοιπο στην Ιταλία 3%. Από τη στιγμή λοιπόν που ορίζονται οι ποσοστώσεις αυτές, για τα συνολικά δηλαδή, για τους ε, συνολικές αυτές ποσοστώσεις για την περιοχή, Υπάρχουν, σύμφωνα με τον κανονισμό που συζητήσαμε και σήμερα το πρωί, υποχρέωση ενημέρωση στην Επιτροπή μηνιαία, κάθε 15 του μηνός δηλαδή, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή τα στοιχεία όσον αφορά την αλληλευτική τους δραστηριότητα. Και θα πρέπει επίσης να δίνουν και μια διορθωτική εγγραφή μετά από διασταύρωση των στοιχείων. Εάν στο τέλος του έτους, γιατί πρόκειται για ποσοστώσεις ετήσιες, υπάρχει απόδειξη ότι τα ποσοστά αυτά ήταν υπερβολικά, ορίζεται ότι μπορεί να υπάρξει μία, ένας μηχανισμός ε, αποζημίωσης αυτό ουσιαστικά κάθε χρόνο γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει δύο τέτοιους μηχανισμούς μείωσης των ποσοστώσεων, έτσι ώστε να υπάρξει τήρηση των κανόνων και να μην ξεπεραστεί το συνολικό ποσό όπως ορίζεται στην αρχή του έτους από τις ποσοστώσεις. Αυτό ισχύει για όλα τα αποθέματα. Τώρα όσον αφορά τον κινητήρινο πτεροτόνο, το 2017 σύμφωνα με τον κανονισμό Δραστηριοποιήθηκε ο μηχανισμός αυτός ε, βάσει τον, του οποίου έπρεπε να ορίζονται οι ποσοστώσεις για τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μόνο εμπλεκόμενο μέρος, συμβαλόμενο μέρος στο IUTC, που ουσιαστικά υιοθέτησε αυτούς τους διαρθωτικούς μηχανισμούς και αυτό το ε, σύστημα αποζημιώσεων ε, θα το λέγαμε. Είναι δηλαδή το μόνο συμβαλόμενο μέρος ε, που για όλα τα αποθέματα υιοθέτησε τέτοιου είδους διοθροτικό μηχανισμό. Όσον αφορά την Ισπανία, τα στοιχεία που υπέβαλε έδειχναν υπεραλίευση 2.465.000 τόνων. Συγγνώμη. 2.465.000 τόνους το 17 αυτό ουσιαστικά αφαιρέθηκε και έγινε καταμερισμός μεταξύ 18 και 19. Για τη Γαλλία για το 17 το ποσοστό ξεπεράστηκε κατά 5.429 τόνους και αυτό το ποσό της υπεραλίευσης έχει κατανεμηθεί για το 2018 και το 2019. Η έλεγχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ε, αξιολόγηση των στοιχείων για αυτά τα είδη του τροπικού τόνου. Εξετάζουμε λοιπόν για το 18 όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που μας έχουν υποβληθεί και το ίδιο θα γίνει και για το 2019. Μέχρι το, το 2018 δεν έχει παρουσιαστεί υπεραλίευση σε κανένα είδος και από καμία χώρα μία σειρά διορθωτικών ε, δράσεων για να ανταποκριθούμε σε αυτή την υπεραλίευση. Έχουν επίσης υιοθετηθεί και από τις εθνικές αρχές. Η Ισπανία έχει θεσπίσει κυρώσεις κατά των αλλιευτικών σκαφών της Ισπανίας. Οι ισπανικές ε, αρχές επίσης έχουν αυξήσει τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, μια νέα ομάδα επιθεωρητών οι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο για καλύτερο έλεγχο των ε, εκφορτώσεων. Δύο λόγια για το IUTC. Αν με επιτρέπετε να μιλήσω και για τον IOTC, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειωθούν τα λιεύματα του κυτρινόπτερου τόνου στον Ειδικό Κενό και ότι θα πρέπει εδώ πέρα να συμμορφωθούμε του σχετικού κανόνε. Θεωρούμε ότι το ψήφισμα του IOTC που εφαρμόστηκε το 2019 δεν το 2018, με συγχωρείτε, δεν μας επιτρέπει να πετύχουμε τα ευκταία αποτελέσματα. Τώρα, για ποιο λόγο είχαμε κάποια αλλιεύματα και κάποιους στόλους που έπρεπε να συμμορφωθούν με συγκεκριμένες μειώσεις αλλιευμάτων, ενώ δεν υπήρχαν οι ίδιοι κανόνες για τα υπόλοιπα συμβαλόμενα μέρη. Ενώ είχαμε και αυξήσεις ε, για τα λιεύματα, για κάποια συμβαλόμενα μέρη τα οποία θεωρητικά έπρεπε να μειώσουν και αυτά τα λιεύματά τους. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά αλλιεύματα του IOTC αυξήθηκαν κατά 3% για το κεντρινόπτερο τόνο σε σχέση με τα επίπεδα του 2014, αντί να μειωθούν δηλαδή. Επίσης, το ψήφισμα του 2018 δεν περίχε κανένα μηχανισμό προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις για την περίπτωση της υπέρβασης των ποσοστώσεων, μόλον ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό. Γι' αυτό το λόγο, φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια τη Επιτροπή Διαχείριση Αλία Τόνου του Ινδικού Ωκεανού, υπέβαλε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη βιώσιμη διαχείριση του κυτρινόπτερου τόνου που αν εφαρμοζόταν θα είχε οδηγήσει σε μια μείωση της τάξης του 12% όσον αφορά τα συνολικά αλλιεύματα κυτρινόπτερου τόνου στον Ειδικό ωκεανό και θα είχε καλύψει όλους τους τόλους και όλους τους ελευτικούς εξοπλισμούς. Δυστυχώς όμως, διότι υπήρχε μια έντονη αντίθεση από τα περισσότερα παράκτια κράτη, που δεν θέλανε να μειωθούν οι δυνατότητε αλίευση των στόλων του. Δεν εγκρίθηκε η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρειάστηκε να συμφωνήσουμε και εμεί με ένα κείμενο το οποίο ήταν λιγότερο φιλόδοξο, το οποίο εν τέλει εγκρίθηκε και που θα οδηγήσει σε μία μείωση μόνο τη τάξη του 7% όσον αφορά τα συνολικά λιεύματα. Τα θετικά όμω νέα είναι ότι εν τέλει ο μηχανισμό αποζημίωση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρήθηκε και επομένως θα εφαρμοστεί από φέτος και στα πλαίσια του IOTC. Τώρα ένα άλλο στοιχείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασκήσει πίεση και συνεχίζει να ασκεί πίεση προκειμένου να έχει μια καλύτερη κάλυψη ελέγχου και παρακολούθησης στα πλαίσια των περιφερειακών αυτών οργανισμών αλληλεία και στα πλαίσια του IOTC και γι' αυτό το λόγο Φέτο εμεί προτείναμε να αυξηθεί αυτή η κάλυψη παρατήρηση σε ένα επίπεδο 100%, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα 50% των στόλων της επί των οποίων υπάρχουν παρατηρητές. Η δική μας η πρόταση δεν έγινε δεχτή από τα, δεχτή από τα υπόλοιπα παράκτια κράτη, επομένως συνεχίζουμε να έχουμε την κάλυψη αυτή ε, με την παρουσία παρατηρητών κατά τρόπο εθελούσιο, αλλά δεν καταφέραμε να πετύχουμε συνένεση, σύμφωνη γνώμη μάλλον με τη δική μας την πρόταση. Ελπίζω ότι τα στοιχεία αυτά σας βοηθούν να καταλάβετε περισσότερο πώς έχει η κατάσταση στα πλαίσια του IOTC και σε σχέση με τι προσπάθειε που έχει καταβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του οργανισμού αυτού και ποιε δυσκολίε έχει αντιμετωπίσει, είναι σημαντικό όμω να καταλάβετε επίση και πώ αναλαμβάνουμε δράση κάθε φορά που προβαίνει σε υπεραλίευση ένα κράτο μέλο, ιδίω όσον αφορά τον κυτρινόπτερο τόνο στον Ινδικό ωκεανό. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε. Η κυρία Ρούση έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την έκθεση σας αυτή. Αναφερθήκατε στην υπεραλίευση από πλευρά ισπανικού των ε, στόλου. Είδαμε ότι ο Μπακαλιάρο όντω υποφέρει πάρα πολύ εξαιτία των δράσεων αυτών του ισπανικού στόλου. Έχετε επιβάλει κάποιες κυρώσει από ό,τι ακούσαμε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες αποκλήσει. το 2017 η Ισπανία έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία στην IOTC στην Επιτροπή Διαχείριση Αλληλεία του Τόνου του Ινδικού Ωκεανού, αριθμητικά δεδομένα τα οποία υπερβαίνουν τα στοιχεία αυτά τα οποία χρησιμοποιήσατε εσεί για να υπολογίσετε τι κυρώσει τα πρόστιμα. Βλέπουμε εκ νέου ότι για το επόμενο έτος υπήρχε υπεραλευίεση από πλευρά τη Ισπανία. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει, προκειμένου τουλάχιστον του χρόνου να αποφύγουμε φαινόμενα υπεραλίευση από την Ισπανία. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε το πρόστιμο σε ποσά σε αριθμητικά δεδομένα τα οποία ήταν τελικά χαμηλότερα από τα πραγματικά αριθματικά δεδομένα. Πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει διορθωτικά μέτρα προκειμένου να ανακατανείμει ποσοστά χαμηλότερα αυτή τη στιγμή στην Ισπανία για του χρόνου. Μιλήσατε επίσης για ένα μηχανισμό αποζημίωσης. Πώς έλαβε χώρο ο μηχανισμός αυτός για την Ισπανία συγκεκριμένα. Πολλές ερωτήσεις που ακούσαμε από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στα αριθμητικά δεδομένα που δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μία πλευρά και από την άλλη Επιτροπή διαχείριση Αλία του Τόνου του Ινδικού Ωκεανού. Αναφερθήκατε σε ένα 59% για την Ισπανία και 39% για την Γαλλία και το υπόλοιπο ποσοστό αντιστοιχεί στην Ιταλία, κάτι τέτοιο είπατε. Ίσως θα έπρεπε να μας πείτε όμως και πόσο σημαντική είναι η αλληλευτική προσπάθεια της Ιταλίας, πιο συγκεκριμένα δηλαδή, με συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα. Ευχαριστώ. Ας δούμε πρώτα τις ερωτήσεις ε, που έχουν υποβληθεί ήδη. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ε, ε, στην IOTC υποβάλλονται πολλά διαφορετικά στοιχεία. Άλλα υποβάλλονται για λόγους επιστημονικούς, για την επιστημονική αξιολόγηση του αποθέματος. Και άλλωστε αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιφερειακές δομές διαχείρισης. Ε, εάν δει κανεί λοιπόν τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται και χρησιμοποιούνται από τους ε, ε, επιστήμονες για να αξιολογηθεί το απόθεμα, δεν είναι ε, απαραίτητα τα στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς ε, σαν ε, Κομισιόν ως αποτέλεσμα των κανόνων ελέγχου. Αυτά είναι στοιχεία δεδομένα τα οποία προκύπτουν από πολλά υποχρεωτικά έγγραφα. Πρώτα απ' όλα έχει κανείς τις αξιολογήσεις από τον καπετάνιο στο ε, logbook στο, στο βιβλίο καταστρώματος. Δεύτερον, στοιχεία από τις εκφορτώσεις μετά από τη ζήγηση. Επίσης, στοιχεία τα οποία προκύπτουν από εκθέσεις επιθεώρησης γιατί μπορεί να υπάρξουν και διαστάσεις ε, όσον αφορά, δηλαδή διαφορές ε, και επομένως σε περίπτωση διαφοράς ε, επιθεώρησης και δηλωμένης εκφόρτωσης τότε υπάρχει διαδικασία παράβασης και επομένως κυρώσεις για τον καπετάνιο. Άρα πρέπει να στέλνουν σωστά στοιχεία. Δεύτερον, Υπάρχουν αξιολογήσεις που γίνονται, εκτιμήσεις που γίνονται από τους επιστήμονες που χρησιμοποιούν πολύ περίπλοκα εργαλεία, ε, εκ των υστέρων ε, ε, υπολογισμούς κλπ. Σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δύσκολο να καταλάβουμε τις διαφορές και ξεκινήσαμε κατά κάποιο τρόπο μια εσωτερική διερεύνηση ε, με μέλη της διοίκησης αλλά και ε, της επιστημονικής ομάδας για να καταλάβουμε καλύτερα τα πράγματα. Όταν όμως μιλάμε για κατανάλωση ποσοστών, ε, ποσοστώσεων πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε στον κανονισμό ελέγχου και βεβαίως αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό για, την αλλιευτική, για τις αλλιευτικές ε, ευκαιρίες βάσει των ποσοστώσεων. Τώρα, όσον αφορά τον νέο ε, κανονισμό ελέγχου, ε, νομίζω από ό,τι μου λέει και ο ότι θα έχουμε τις ίδιες αξίες. Δηλαδή θα υπάρχει ένα rollover των αξιών που ανέφερα, των τιμών που ανέφερα προηγουμένως όπου ε, θα προσθεθούν όλες οι μειώσεις ε, που ε, ενδεχομένως θα καταστεί απαραίτητο να εφαρμοστούν τα κράτη-μέλη, εάν υπάρχει οποιαδήποτε μείωση. Έγινε λόγος για έναν πολλαπλασιαστικό παράγοντα. Είναι γεγονός ότι ο κανονισμός ελέγχου προβλέπει κατά κάποιο τρόπο μία επιπλέον κύρωση και αντίστοιχη μείωση της αλλιευτικής ε, ε, ικανότητας, αλλά αυτό μπορεί να συμβαίνει εάν ε, η διαφορά ξεπερνάει το 10%. Αλλά εδώ δεν είχαμε τέτοια περίπτωση, ήταν λιγότερο από 10% της διαθέσιμη, του διαθέσιμου ΤΑΚ. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αυτός ο μηχανισμός μείωσης υπάρχει από δημιουργίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία κατεστική απρακτική και είχαμε πάντα στην ε, ομάδα διαχείρισης των δεδομένων συναδέλφους που μπορούσαν να ελέγξουν ε, το, το, τους, ε, τις εκθέσεις αναχώρα και επομένως τα ΤΑΚ και επομένως να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις. Έγινε και μια ερώτηση από τον Πρόεδρο όσον αφορά την... um, την κατανομή των ε, στοιχείων, ναι, ε, έχουμε 14 με ισπανική σημαία, 12 με γαλλική και ένα με άλλη σημαία. Τι είπατε, κάτι αναφέρατε στη διαδικασία payback, αποζημίωσης, επιστροφής. Δεν έχει ξεκινήσει τώρα, θα ξεκινήσει. Καταβολή των χρημάτων. Η διαδικασία payback είναι δύο φορές το χρόνο. Δύο φορές το χρόνο λοιπόν γίνονται οι πληρωμές όταν έχουμε πλέον τα τελικά στοιχεία για το 2018 για το κυτρινόπτερο δεν έχουμε ε, στοιχεία υπεραλίευσης άρα προς ώρας δεν ε, υπάρχει payback το payback στο οποίο, το οποίο έχει ήδη λάβει χώρα αφορά το 2017. Έχουμε επίσης μείωση των ποσοστώσεων για την Ισπανία και το 18 και το 19. Ωραία, ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι δεν απαντήσατε ε, λέει η κυρία Ρόζ, σχετικά ε, με το πώς θα, ε, τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρετε να απαγορεύσετε, να αποτρέψετε την Ισπανία να ξαναψαρέψει. Πρώτον, το ίδιο το κράτος μέλος έχει αυτή την ευθύνη, δηλαδή θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν ξεπερνούν, δεν παραβιάζουν τις ποσοστώσεις και αυτός ο μηχανισμός επιστροφής, payback, είναι αποτρεπτικός για τα κράτη. Τώρα, όσον αφορά την Ισπανία. Η Ισπανία έχει εφαρμόσει ήδη από το 2018 ε, συμπληρωματικά μέτρα. Το 2017 δεν ε, ε, τους είχαν δοθεί συγκεκριμένη ποσόστοση ανασκάφος. Επομένως δεν είχε γίνει κατανομή ανασκάφος. Από το 2018 η Ισπανία έχει ε, κατανείμει συγκεκριμένες ποσοστώσεις ανασκάφος, άρα ε, μπορεί να ολοκληρωθεί καλύτερα, να εφαρμοστεί καλύτερη διαδικασία επιτήρησης ε, και ελέγχου. Είναι ένα καλό μέτρο. Επιπροσθέτως, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να πω ότι η Ισπανία έχει ενισχύσει τις διαδικασίες ελέγχου στον στόλο της πρώτον προβλέπουν συγκεκριμένες κυρώσεις για όσους έχουν ξεπεράσει το, την ποσόστοσή τους. Επίσης, ε, έρχονται σε επαφή με τις Σεϊχέλες που είναι η κύρια χώρα στην οποία γίνεται εκφόρτωση του ε, κυτρινόπτερου, έτσι ώστε να ελέγχουν τους, ε, τις εκφορτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του ελόγου όσον αφορά τώρα εκφορτώσεις τρίτων χωρών στην ουσία εξαρτόμαστε 100% στον, ε, στην ικανότητα ελέγχου ε, ε, της συγκεκριμένης χώρας. Πέστε μας και κάτι για το μέλλον πριν κλείσουμε το θέμα. 21% μονάχα του, του τόνου του Ινδικού ωκεανού αλλιεύουμε. Ξέρουμε τα τονάζ. Ξέρουμε τι, τους, τις ελιευμένες ποσότητες, ξέρουμε λίγο οι άλλοι τι ψαρεύουν, ποιες είναι οι ποσότητες δηλαδή ελιευμένες. Ε, μπορεί να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Ε, μας είπατε βέβαια ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες ε, δεν θέλουν, αντιδρούν στους ελέγχους και υπάρχουν χώρες οι οποίες αλλιεύουν αυτή τη στιγμή πολύ στον Ειδικό ωκεανό. Ας πούμε, η περίπτωση της Ινδίας. Εκεί επιτρέπεται την υπεραλίευση σε μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός ε, διαρκώς ε, αυξάνεται και επομένως λογικά πιέζονται τα πλέτα αποθέματα. Αλλά μία, δύο, τρεις, πόσες φορές θα το επιτρέπετε. Θα ζητήσω όμως ε, την βοήθεια εδώ της συναδέλφου που είναι επικεφαλής της ΑΕΤΣΗ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την ερώτησή σας, γιατί είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Η απάντηση πάντως δεν είναι εύκολη. Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό που μας λέτε. Ήταν ε, προβληματισμός μας ε, και, και δικός μας λοιπόν στις διαπραγματεύσεις πέρα από όλα αυτά που αναφέρθηκε προηγουμένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Εξακολουθεί να υπάρχει το θέμα ε, της διαχείρισης των αποθεμάτων στον Ειδικό ωκεανό και βλέπουμε πραγματικά πολύ μεγάλη αντίσταση. Πολλές χώρες ζητούν ε, από τις γειτονικές ε, χώρες ε, να κάνουν, να καταβάλουν κάποια προσπάθεια. Αλλά μην λησμονούμε ότι οι ωκεανοί είναι ενιαίοι, τα βαθαία ύδατα επίσης, τα πελαγικά είδη ε, το ίδιο άρα θα πρέπει να βρούμε συνολικά το πρόβλημα, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες ε, των αναπτυσσομένων χωρών. Ε, δηλαδή η προσπάθεια συντήρησης αποθεμάτων δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς ίδιο, ίδια από όλες τις χώρες. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να καταλάβουν όλες τις χώρες αιτησία ότι πρέπει να κάνουν κάτι. Πέρα από τις πρωτοβουλίες που έχουμε και την επαφή με άλλες χώρες IOTC που έχουν ε, ενταθεί, υποστηρίζουμε και κάποιες, υποσ... κάποιες ε, πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους συναδέλφους ε, της ανάπτυξης ε, και με δικιά μας ε, χρηματοδότηση, έτσι ώστε να βοηθήσουμε κάποιες χώρες της περιοχής όσον αφορά την συλλογή δεδομένων, γιατί έχουμε προβλήματα και για τον Ειδικό ωκεανό. Πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται, πώς πρέπει να γίνεται σωστότερα η διαχείριση και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε επιστημονικά στοιχεία γι' αυτό γιατί διαφορετικά θα αποδεκατιστεί ο τόνος και ο κιτρινόπτερος και δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε την ε, αλία. Επομένως, βοηθάμε τις χώρες αυτές, οργανώνουμε εργαστήρια, workshops. Θέλουμε να ε, βάλουμε όλες τις χώρες ε, σε αυτήν την διαδικασία αξιολόγησης και προσπάθειας, αλλά βεβαίως υπάρχουν αντιστάσεις και δεν ξέρω αν απήντησα με αυτά τα λίγα λόγια σε αυτό που ρωτήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε Κομισιόν. Πολύ υποβοηθητική, καθώς επίσης και ενδιαφέρουσα ε, και πλήρης η απάντησή σας. Επόμενο θέμα. 15 και 16 πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή τη Συμφωνία Ελευτική Σύμπραξη μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη Δημοκρατία τη Γουινέα Μπισάου. Να σα υπενθυμίσω ότι πρόκειται για ένα πρωτοκόλλο το οποίο υπεγράφει και άρχισε να εφαρμόζεται από τον Ιούνιο για μια περίοδο 5 ετών. Εμείς ε, συμβάλλουμε κατά 15,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα τέσσερα δίνονται για την πρόθεση του τομέα της αλίας της Γουινέας Μπισάου. Η Γωνία Μπισάου είναι από τις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη και έχει ένα αναλυτικό τομέα ο οποίος είναι υποαναπτυγμένος αυτή τη στιγμή. Επομένω, σαφώς υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φεραίρα, ο οποίος όμως αποσιάζει, αν ήταν πάντως παρόν, θα του έλεγα ότι η έκθεσή του είναι ιδιαίτερα διεξοδική, πάρα πολύ καλή, αλλά έχουμε την κυρία Περέρα που θα τον αντικαταστήσει. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, ο Ζωάν Φιρέρα σας ζητά συγγνώμη που δεν είσαι θέση να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση. Θα κάνω εγώ στη θέση του μια σύντομη παρουσίαση του σχεδίου σύστασης, καθώς επίσης και του σχεδίου έκθεσης του μήνυμα Θετικού ψηφίσματος. Η πρώτη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση χρονολογείται από το 1980. Έκτοτε έχουν συναυθεί διάφορα πρωτόκολλα τα οποία έτυχαν διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιο πρόσφατο πρωτόκολλο αναγνωρίζει την ανάγκη επικαιροποίησης των δεδομένων που έχουμε όσον αφορά την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον τομέα λίας της Δημοκρατίας της βουινεα Μπισάου. Το εφιστάμενο πρωτόκολλο βασίζεται σε μια συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλίας για την περίοδο μέχρι το 2024 που θα αρχίσει να ισχύει προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής, δηλαδή 15 Νοεμβρίου 2018. Κατά αυτόν τον τρόπο, σκάφη από πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα λευτικά ύδατα της Γουινέας Μπισάου για τις ακόλουθες κατηγορίες. Μηχανότρατες γαρίδας με ψυκτικές εγκαταστάσεις, μηχανότρατες για κεφαλόποδα και για την αλία ηχθείων με ψυκτικές εγκαταστάσεις, μηχανότρατες αλίες μικρών πελαγικών ειδών και θυναλιευτικά με ψυκτικές εγκαταστάσεις και παραγαδιάρικα, καθώς επίσης και για θυναλιευτικά με καλάμι. Στις πρώτες τρεις κατηγορίες προβλέπεται μεγαλύτερη χρονική περίοδος από ό,τι στις δύο τελευταίες. Υπάρχουν, ε, όπως σας είπα, πολλές κατηγορίες αλληλευτικών ειδών που καλύπτονται από τη συμφωνία αυτή και από το μετέπειτα πρωτόκολλο και έχουμε ανάμεσα κατηγορίες αυτές αλληλευτικών ειδών τον τόνο, διάφορα θηνοειδή, γαρίδες και διάφορα κεφαλόποδα. Έχουμε επίση μια συγκεκριμένη σύσταση τη ICAT, η οποία θα πρέπει και αυτή με τη σειρά τη να εφαρμοστεί στα πλαίσια του πρωτοκόλλου αυτού. Ο εισηγητή, ο συντάκτη γνωμοδότηση θεωρεί ότι θα πρέπει να εγκριθεί το πρωτόκολλο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ίδια την Γουινέα Μπισάου και τον δευτικό τη κλάδο, αλλά και για τα λευτικά σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη δική του τη βιωσιμότητα. Θα γίνει μάλιστα και μια πολύ λεπτομεριακή αξιολόγηση του πρωτοκόλλου αυτού, καθώ επίση και τη εφαρμογή του σε μερικά χρόνια. Έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να υποβάλουμε αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο σύστασης καθώς επίσης και ένα μη νομοθετικό ψήφισμα που θα εκφράζει την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύω της συμφωνίας αυτής και για την πενταετή δηλαδή περίοδο. Θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση η συμφωνία αυτή θα πρέπει να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη του λευτικού κλάδου της δημοκρατίας του, της Γουινέας Μπισάου και βέβαια θα πρέπει να προωθήσει και τους παρενθερείς κλάδους που εξαρτώνται δηλαδή από την αλία και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η συμφωνία αυτή να προωθήσει την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλευτικών πόρων της χώρας αυτής. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, αλλά και μέσω άλλων ευρωπαϊκών εργαλείων όλη την απαραίτητη χρηματοδότηση, προκειμένου να καταφέρουμε να συνεργαστούμε περισσότερο με τη χώρα αυτή σε διεθνές αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του EDF, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και για τη βελτίωση των ελευτικών υποδομών, για την καλύτερη ανάπτυξη ελευτικών πόρων και για την καλύτερη ανάπτυξη των απαραίτητων εξοπλισμών εκφόρτωσης και μεταπίεσης επεξεργασίας των θαλασσινών και των υπολοιπών αλλιευτικών ειδών. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε καλύτερου τρόπου για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή απορρόφηση των πόρων αυτών από την Γουινέα Μπισάου. Πρόσφατα είδαμε ότι η απορρόφηση αυτή δεν ήταν επαρκή και θα πρέπει να, γίνουν περισσότερε προσπάθειε προκειμένου να απορροφώνται τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά και να έχουμε και θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τον αλλιευτικό κλάδο τη Γουινέα Μπισάου. Βέβαια, παράλληλα χρειαζόμαστε και περισσότερα στατιστικά δεδομένα από τη χώρα αυτή, προκειμένου να μπορούμε και εμεί να παρακολουθούμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση του αλλιευτικού κλάδου. Θεωρώ ότι μπορούμε μέσω της συμφωνίας αυτής και με το πρωτόκολλο αυτό να βοηθήσουμε την Γουινέα Μπισάο για τον αλλιευτικό της κλάδο και να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να καταρτίζει καλύτερα στατιστικά δεδομένα όσον αφορά τον ελευτικό κλάδο. Πρέπει λοιπόν να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συμφωνία αυτή και μέσω της συμφωνίας αυτής θα καταφέρουμε επίσης να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της α, άναρχης αδήλωτης αλίας και ελπίζω ότι από το Φεβρουάριο του 2020 και μετά ως Επιτροπή Αλίας θα μπορέσουμε να μεταβούμε επί τόπου για να έχουμε και εμείς ως μέλη της Επιτροπής αυτής μια καλύτερη, πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα στον αφορά τον ελευτικό κλάδο της χώρας αυτής. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό επίσης να ε, συμμετέχουν στην επίσκεψη αυτή, στην αποστολή μας αυτή και συνάδελφοι και από άλλες επιτροπές. Όντω, το Φεβρουάριο θα λάβει χώρα η επίσκεψη αυτή, λέει ο Πρόεδρο. Ο κύριο Μπέρκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρόν. Δεν νομίζω. Είναι καθοδόν, μάλιστα. Λοιπόν, εφόσον είναι καθοδόν, τότε ας περιμένουμε να έρθει για να συνεχίσουμε την εξέταση του σημείου αυτού. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να πάρουν το λόγο συνάδελφοι. Ίσως να αναστείλουμε την εξέταση του σημείου αυτού και να επανέλθουμε λίγο αργότερα όταν έρθει και ο αρμόδιος πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ακούσει τις παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν οι ευρωβουλευτές, έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Μήπως να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Μπαρτόλο για το επόμενο σημείο αλλά και πάλι ας δούμε αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μπορούσε να σας απαντήσει. Μάλλον ο κύριος Ντεμπλίκ, ο κύριος Νούντς είναι παρόντες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, για όλα τα αναπομείνοντα σημεία τη μερίσια διάταξη έχουμε ανάγκη από του ίδιου εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι δεν είναι παρόντε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να έρθουν κάποια στιγμή προκειμένου να μπορέσουμε να αναλύσουμε τα σημεία αυτά στη μερίσια διάταξη. Δεν είναι καθόλου θετικό βέβαια το ότι δεν είναι παρόντε μας λέτε ότι είναι καθοδόν. Απευθύνομαι στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι στην αίθουσα. Τι ακριβώς εννοείτε, σε πόση ώρα. This is what mobile phones are for. You can't use them on fishing boats, according to Mrs. Mummery, but uh, you can at least use them to try and find the Commission. Να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τον αρμόδιο υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δείτε, σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση πριν τις 6.30. Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή ένα δεκάλεπτο διάλειμμα.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 Okay, start again. Thank you, Mr. for uh, joining us. Uh, we've had a presentation. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε, είχαμε μια ε, εκπρόσωπο του εισηγητού, ο οποίος, η οποία μάλλον μας παρουσίασε την έκθεση του εισηγητού. Um, by Mr. Ferreira. Um... Η παρουσίαση έγινε από την κυρία Φερέρα. Ακούστηκαν και κάποια σχόλια Μάλλον θα ακούσουμε και κάποια σχόλια. Ο κύριος Γκονζάλης Κασάρες. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε, Πρόεδρε. Η ανανέωση αυτού του, της Αλληλευτικής Συμφωνίας ε, είναι πολύ καλοδεχούμενη, κυρίως ε, για τα 16 πλοία της Γαλλικής από τα 24 της Ισπανίας που ψαρεύουν στην Γουινέα Ισάου είχαμε μεγάλη ανησυχία λόγω της συμφωνίας με το Μαρόκο ε, και εδώ τουλάχιστον βλέπουμε ότι στην περίπτωση της ε, Γουινέας Μπισάου έχουμε μία από τις τρεις ε, συμφωνίες μικτής αλίας και αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης η συμφωνία αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού, βελτιώνει επίσης ε, την ε, ε, οικονομική κατάσταση του τοπικού κλάδου. Και επίσης και για τη δική μας περίπτωση έχουμε η υποστήριξη του κλάδου. Το θέμα είναι να δούμε πόσα, πόσοι είναι, θα είναι οι αλληλείς της Γουινέας που θα εργαστούν στον Ευρωπαϊκό Στόλο. Επίσης, θα πρέπει να ε, ε, ξεπεραστεί το πρόβλημα ε, της μη συμμόρφωσης με υγειονομικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει αναστολή των εξαγωγών από τη χώρα αυτή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά λόγω έλλειψης εργαστηρίων ανάλυσης κτλ. Αυτό θα πρέπει να ξεπεραστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι γεγονός ότι εμείς θα προβλέψουμε και μία αποστολή στη Γουινέα για να δούμε τα πράγματα από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κομισιόν γιατί έχει ολοκληρώσει συμφωνίε όπως αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερέρα. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί έκανε εξαιρετική εργασία. Ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, όσον αφορά ε, τα αλληλευτικά εργαλεία τρίτων χωρών. Αναφέρομαι κυρίως σε ασιατικούς στόλους. Εκτιμούμε ότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω. Η έκθεση μάλιστα αναφέρει ήδη ότι θα πρέπει να γίνουν ε, σχετικές ε, ε, μελέτες. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι πόροι που θα δοθούν στον κλάδο αυτό. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη είναι τις ε, τοπικές οργανώσεις αλλιέων που θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να έχουμε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Η κυρία Τόμασιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Υποστηρίζω τη συμφωνία αυτή διότι ε, συμπεριλαμβάνει και το σκέλος της καταπολέμησης ε, της ε, ε παράνομης αλίας και επίσης δίνεται και βοήθεια σε τοπικούς ψαράδες. Ευχαριστώ κύριος Βαντέλεν. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω, λέει ο κύριος Βαντάλεν, ε, την, ε, τον εισηγητή για αυτήν την εξαιρετική έκθεση που μας έχει υποβάλει. Είμαστε υπέρ του κειμένου, το οποίο θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά ισορροπημένο. Όμως, η κατάσταση στη Γουινέα Μπισάου είναι πάρα πολύ περίπλοκη τούτη τη στιγμή. Την 8η Νοεμβρίου ο, παρετήθηκε ο Πρωθυπουργός Υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις στη χώρα και την, ε, στις 14 Νοεμβρίου θα γίνουν ε, προεδρικές εκλογές. Η κατάσταση λοιπόν είναι ασταθής. Η Κομισιόν θα μπορούσε να μας πει εάν αυτό έχει και ποια επίπτωση κυρίως στην ε, Αλία, γιατί η Αλία αντιπροσωπεύει 4% του ΑΕΠ. Τούτων λεχθέντων, στα πλαίσια ενός ψηφίσματος, ίσως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, και οι δραστηριότητες ε, των κινέζικων πλοίων ε, στον κόλπο, στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου. Οι Κινέζοι ψαρεύουν πολύ, μετατρέπουν, μεταποιούν το αλίευμα ε, σε ε, ε, άλευρα και επομένως ρωτώ την Κομισιόν μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να σταματήσουν αυτές οι δραστηριότητες της Κίνας. Η Κίνα η οποία δεν ψαρεύει με βιώσιμο τρόπο και που στην ουσία θέλει μονάχα να εξάγει, να μετατρέπει, συγγνώμη, να μεταποιεί σε άλευρα και σε έλεα αλλά αυτό όμως σημαίνει ότι θέτει σε κίνδυνο ε, τις, ε, αλλιε... τους αλλιευτικούς πόρους. Νομίζω ότι με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αναλύσουμε αυτήν την ε, κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρόντ. Ε, ζήτησα το λόγο γιατί είμαι η συγγήτρια από την Κομισιόν ΔΕΒΕ για τις συμφωνίες με την Γουινέα Μπισάου. Στην γνωμοδότησή μου ζήτησα να συμπεριληφθούν κάποια στοιχεία. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική της αλίας θα πρέπει να είναι συνεκτική με τους αναπτυξιακούς στόχους. Ε, επίσης, η πρόσβαση του ευρωπαϊκού στόλου δεν θα πρέπει να ε, διασαλεύσει την ε, ασφάλεια, επισητιστική ασφάλεια των τοπικών πληθυσμών. Ζήτησε επίσης πλήρη διαφάνεια της χρήσης των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσίευση πλήρους καταλόγου των ε, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων και, και ε, επίσκεψη επιτόπου αντιπροσωπείας. Πιστεύω επίσης ε, ότι είναι σημαντικό να τίνουμε νευρικόνους και να φουγκραζόμαστε τις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε εδώ εκπροσώπους της χώρας, τους συναντήσαμε με την κυρία Σάλιβαν, μιλήσαμε για τον ρόλο της γυναίκας που πρέπει, στην Αλία που πρέπει να ληφθεί υπόψη, τον ρόλο της τοπικής ψυχικής το, το, το, το, κομμάτι της αυτοσυτιστικής ε, ε, αλληλείας που είναι πολύ σημαντικό για την χώρα αυτή. Αυτά ήθελα και δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βερνά. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίγα. Πρόκειται εδώ για μια συμφωνία που είναι σημαντική ε, για, την, ε, για τον αλληλευτικό τομέα της Ισπανίας και της χώρας των Βάσκων ε, ιδιαιτέρως. Θέλω να πω τα εξής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δυνατότητες αλληλείας τα τρία τελευταία χρόνια ε, βασίστηκαν ε, στα ε, ΤΑΚ και νομίζω ότι είναι μεγάλη πρόκληση το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου όντως και δεν θέλω να το επαναλάβω πραγματικά, αλλά το είπαμε και σε κάθε παρόμοια συζήτηση ε, για τέτοιου είδους συμφωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικό η ανάπτυξη του τοπικού ε, κλάδου ή η τοπική ανάπτυξη του κλάδου αν θέλετε είναι πάρα πολύ σημαντικό θα πρέπει να αναπτυχθεί ο κλάδος στη Γουινέα Μπισάου ε, όσον αφορά τώρα τους ε, ναυτικούς ε, που θα προσληφθούν και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Οι επενδύσεις ε, από πλευράς των κρατών μελών είναι πολύ σημαντικές έτσι ώστε να σταματήσει πια αυτή η ανισορροπία. Ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν το εξής. Όταν μιλάμε για τοπική ανάπτυξη ε, μπορούμε να έχουμε κάποια ε, συγκεκριμένα προγράμματα, να μας πει ποιοι, κάποια προγράμματα τα οποία ε, είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνική κατάσταση, κυρίως δε εξειδικευμένα προγράμματα για την ανάπτυξη της θέσης της γυναίκας στον τομέα της αλίας, εάν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα και τι σκοπεύουν, αν υπάρχει πρόθεση να γίνει κάτι στο μέλλον. Να στραφώ προς την Επιτροπή. Προσέξα. Είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε την έξι χιλιάς Φερέρα. Γιατί συνειδητοποιώ ότι εδώ ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι περιορισμένος. Αλλά πρόκειται για μια πολύ καλή πρόταση. Και θα θέλαμε να ξέρουμε αν μπορείτε να απαντήσετε με θετικό τρόπο εδώ, σαν Επιτροπή, σε αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Πρόκειται για μια εξαιρετική άσκηση. Θα στηρίξουμε τις περισσότερες από τις συστάσεις της έκθεσης αυτής. Πρόκειται για μια σημαντική πρόταση και για το στόλο μας, αλλά και για τη χώρα αυτή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Αλία. Μετά από έξι συναντήσεις, ένα γύρο έξι συναντήσεων ε, με τις αρχές της Γουινέας Μπισάου, νομίζω το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Έχουμε αλλάξει κλίμακα. Περισσότερα ήδη, οι όγκοι, οι ποσότητες έχουν αυξηθεί και επίσης σήμερα στηρίζει ο κλάδος και έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για μια πραγματικά βιώσιμη πολιτική αλία στη Γουινέα Βισάου. Πολλές λοιπόν είναι οι προκλήσεις και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε τη συμφωνία αυτή και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης που είναι στην καρδιά της. Μιλήσαμε για την απασχόληση των αλλιέων. Πρόκειται για μια συμφωνία. Αν κοιτάξει κανεί τι διατάξει αυτού του πρωτοκόλλου, διαπιστώνουμε ότι θέλουμε να δούμε τι επιπτώσει επί τη απασχόληση. Τα αλλιευτικά σκάφη, τα ευρωπαϊκά, οι δηλαδή, και οι προτάσεις ε, της συνάντηση της Μικτής Επιτροπής του Οκτωβρίου, αν δείτε τα πρακτικά αυτή της συνεδρίασης, γιατί και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο έχουμε υποβάλει όλα αυτά τα πρακτικά όλων των συναντήσεων που είχαμε. Περίπου 150 αλείς από τη Γουινέα Βισάου εργάζονται στον Ευρωπαϊκό Αλλιευτικό Στόλο. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν λοιπόν επιπτώσεις και στην απασχόληση και στην τοπική ανάπτυξη κάτι που προβλέπεται από όλες αυτές τις προτάσεις και διατάξεις. Έλεγχος της παραγωγής, αυτό είναι για μας μια πάγια θέση. Λάβουμε υπόψη μας όλους τους επιστήμονες πριν καθορίσουμε τις ποσότητες για όλα τα είδη. Έχουμε επίσης και μια μεικτή επιστημονική επιτροπή, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αρχές του 20. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός ότι περνάμε σε ένα σύστημα διαχείρισης με βάση ποσοστώσεις. Μέχρι τώρα βασιζόμασταν στις δυνατότητες αλλιεύσης τονάζ των αλλιευτικών σκαφών και από εκεί και πέρα μπορούσαν να αλλιεύουν ε, κατά το δοκούν. Αυτό όμως το σύστημα έχει τελειώσει. Σήμερα υπάρχει συγκεκριμένη ποσόστοση με συγκεκριμένους αριθμούς και αυτό που ζητήσαμε και από τη Γουινέα Μπισάου είναι και αυτοί να υιοθετήσουν ένα τέτοιο σύστημα διαχείρισης βασιζόμενο σε ποσοστώσεις για το σύνολο των αλληλευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και για τον κινέζικο στόλο και για τον ε, τοπικό. Έχουμε μία συμφωνία εξάλλου μεταξύ Γουινέας Μπισάου και Κίνας. Ίσως να μην είναι τόσο διαφανής όσο η δική μας, η οποία ανανεώνεται αυτή την εποχή. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις και σε αυτό το τομέα. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι ποια είναι η εθνικότητα του ελευτικού σκάφους, αλλά εάν τηρούνται οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων με αυτές που έχουμε επιβάλει στον Ευρωπαϊκό Αλλιευτικό Στόλο. Σχέδιο διαχείρισης των αλλιευμάτων. Κάτι που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δραστηριότητα όλων των, στόλων που βρίσκονται στην περιοχή. 4 εκατομμύρια το χρόνο είναι το ποσό για τη στήριξη του αληφτικού τομέα στη Γουινέα Μπισάου. Κοιτάξτε τα πρακτικά, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης τον Οκτώβριο της Μικτής Επιτροπής, ο προγραμματισμός και μία σειρά συγκεκριμένων μέτρων. Βιώσιμη διαχείριση της αλίας, ενίσχυση του επιστημονικού τομέα, επιτήρηση, έλεγχη και στήριξη στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της α, μικρής κλίμακας ερασιτεχνικής αλίας. Αυτή είναι η στόχη. Ξέρω ότι αυτό που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η στήριξη στην ερασιτεχνική αλία, στην μικρή, μικρής κλίμακας μάλλον αλία. Όσον αφορά τις μικρές μονάδες για την αποξήρανση και την επεξεργασία με καπνό των αλλιευμάτων, καθώς και τη δυνατότητα εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των προϊόντων μεταποιημένων ε, από την Γουινέα Μπισάου. Ήδη εξάγουν προς κάποιες άλλες χώρες. Θα πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση της ε, μονάδας αυτής γιατί θεωρούμε ότι πρέπει πέρα από τη συμφωνία για την αλία να υπάρχει και μια στήριξη όλων αυτών των δραστηριοτήτων που μπορεί να αποφέρουν έσοδα στη χώρα αυτή. Όσον αφορά τα ψαράλευρα, τα ηχθιάλευρα, αυτό είναι ένα πρόβλημα και σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε στη Γουινέα Μπισάου δεν υπάρχει μονάδα παραγωγής τέτοιων ε, προϊόντων που να χρησιμοποιεί ε, φρέσκα ψάρια. Και δεν γνωρίζουμε να υπάρχει σχέδιο για την ε, παραγωγή αυτή επιτόπου. Όπως και η Επιτροπή Ανάπτυξης, θεωρούμε και εμείς ότι πρόκειται για πολύ θετικές διατάξεις όσον αφορά την ε, συμμετοχή σε είδος έτσι ώστε να μπορέσει ένα τμήμα αυτών των ε, προϊόντων της αλίας να απευθύνεται στις τοπικές κοινωνίες αυτοσύτηση. Παρακολουθούμε λοιπόν την εφαρμογή ε, της συμφωνίας από κοινού με τους συναδέλφους που βρίσκονται επί τόπου 24 Νοεμβρίου θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, στηρίζει την κυβέρνηση του Αριστίτ Κομές. Με αυτή την κυβέρνηση έχουμε επαφές. Αυτή εξάλλου είναι η πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να υπάρξουν εκλογές η αληφτική δραστηριότητα εντωμεταξύ συνεχίζει και οι τακτικές μας ε, επαφές με τις αρχές ε, σε εθνικό επίπεδο δεν έχουν επηρεαστεί με κανένα τρόπο από τα πολιτικά γεγονότα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι σαφές ότι ε, ο εισηγητής και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές θέλουν να έχουμε μία θετική εταιρική σχέση με την Γουινέα Μπισάου που όχι μόνο να αποδώσει από επενδυτικής πλευράς αλλά να συμβάλλει τελικά στην καλύτερη κατάσταση της αλίας στην χώρα αυτή. Προτού περάσουμε στο επόμενο σημείο, να σας πω ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 3η 19 Νοεμβρίου, 5 η ώρα το απόγευμα. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης, σύναψη τη συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ. Ο κύριος Μπαρτόλο είναι ο συγητή. Ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βιετνάμ σαφώς δημιουργεί πάρα πολλέ θετικέ ευκαιρίε και για τη χώρα αυτή, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω η χώρα αυτή να μπορεί πραγματικά να ακολουθεί τους κανόνες προκειμένου να μπορούμε τελικά μέσω τη συμφωνίας αυτή ελεύθερων συναλλαγών να καλύψουμε θετικά τον ελευτικό τομέα τόσο του Βιετνάμ όσο και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταφέρουμε να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον. Όπω λέω και στην έκθεσή μου που έχετε ενώπιον σα, είναι πολύ θετικό το ότι η συμφωνία αυτή αναγνωρίζει το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια βιώσιμη διαχείριση των ζώων των θαλάσσιων πόρων, καθώς επίσης και των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δεσμεύσει και από τι δύο πλευρέ για να καταπολεμηθεί η παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλία. Και θεωρώ ότι είναι θετικό αυτή τη στιγμή το ότι η κυβέρνηση του Βιετνάμ ζήτησε να αρχίσει να συμμετέχει στην Επιτροπή Αλίας του Δυτικού και του Κεντρικού Ειρηνικού. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια πιο στενή συνεργασία με τη χώρα αυτή για τα ζητήματα αυτά τα οποία έθιξα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό η κυβέρνηση του Βιετνάμ να ολοκληρώσει την εσωτερική εθνική της νομοθεσία όσον αφορά την μεταρρύθμιση του ελευτικού τομέα είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς συντονισμού, παρακολούθησης και ελέγχου της παράνομης αλίας. Οι πρώτες πρωτοβουλίες κινούνται προς σωστή κατεύθυνση. Στα πλαίσια της καθέ εκθεσής μου θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφαιρθούμε στα βασικά νομοθετικά κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όσον αφορά το Βιετνάμ. Δεν υπάρχει κατάλληλη αυτή τη στιγμή καταγραφή του ελευτικού στόλου καθώς επίσης των ελευτικών προσπαθειών του αληφτικού πληθυσμού, καθώς επίσης και των προσπαθειών που καταβάλει η χώρα ή που θα έπρεπε να καταβάλει για την καταπολέμηση της παράνομης και της αδήλωτης αλίας. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα τα οποία έχει, όπως για παράδειγμα η προδοποίηση με την κίτρινη κάρτα. Αυτό ήδη έγινε τον Οκτώβριο του 2017 θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των πρωτοποιήσεων αυτών να καταφέρει βέβαια να ενθαρρύνει τη χώρα αυτή προκειμένου να μεταρρυθμίσει τον αλλιευτικό της κλάδο. Επίσης, οι προτιμησιακοί δασμοί που προτείνουμε προς το Βιετνάμ θα πρέπει όμως να συνοδεύονται και από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεσμεύσεις της χώρας αυτής. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί εκ του σύνογγης και συστηματικά την κατάσταση, προκειμένου οι ίδιες οι αρχές ρυθμιστικές του Βιετνάμ να αρχίσουν να παρακολουθούν πιο αυστηρά τον ρευτικό του στόλο και να αρχίσουν να επιβάλλουν κυρώσεις ή να εφαρμόζουν κανόνες προκειμένου να ε, γίνονται σωστά και δραστηριότητες αλλήλευσης αλλά και δραστηριότητες εξαγωγής προς ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω επίση ότι θα πρέπει ο ελευτικό κλάδο του Βιετνάμ να αρχίσει να συνάδει περισσότερο με του διεθνεί στόχου βιώσιμη αλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή, στη προκειμένου, όπως και η κίτρινη η κόκκινη κάρτα, προκειμένου να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εισαγωγέ των ηλεκτρικών προϊόντων από το Βιετνάμ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα συνάδουν με του κανόνε και θα καταλήγουμε να έχουμε τελικά ασφαλή προϊόντα για του Ευρωπαίου πολίτε. Σαφώ λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει η συμφωνία αυτή να επικυρωθεί αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιφέρουμε και τις απαραίτητες βελτιώσεις. Είμαι στην διάθεσή σας για τυχόν παρατηρήσεις ή τυχόν ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Από διαδικαστικής πλευράς πρέπει να σας πω ότι καλύπτουμε από κοινού τα σημεία 17 και 18. Έχουμε δηλαδή την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότηση από τη μια πλευρά και του σχεδίου γνωμοδότηση επί της πρότασης ψηφίσματος. Κύριε Μπαρτόλο, Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτή είναι μια γνωμοδότηση που υποβάλλουμε προς την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Αυτή είναι η επιτροπή η οποία βλέπει, αν θέλετε, τη σφαιρική εικόνα τη κατάσταση. Εμεί επικεντρωνόμαστε στην ελευτική πτυχή τη συμφωνία αυτή. Από εμπειρίε όμω ξέρουμε ότι οι καθήλυνα αρμόδιε επιτροπέ δεν λαμβάνουν δεόντω υπόψη τι γνωμοδοτήσει των υπολείπων επιτροπών. Επομένως, μήπως θα έπρεπε να έχουμε μια διατύπωση λίγο πιο αυστηρή σε σχέση με τη χρησιμοποίηση της κίτρινης ή της κόκκινης κάρτας, προκειμένου να στείλουμε όσο το δυνατόν το πιο χειρό μήνυμα προς την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Ας το έχουμε αυτό κατά νου και ας α, ακούσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Σρέιερ Πιέρικ να ευχαριστήσω και τον συντάκτη της εκνομοδότησης. Και να σας πω ότι εγώ προσωπικά συμφωνώ με τον κύριο Μπάρτολο. Η Επιτροπή Ίντα ασχολείται με το θέμα της παράνομης και λαθρέας άναρχης αλίας επιθυμεί να ληφθούν μέτρα για να καταπολεμηθεί αυτού του είδους η λαθρέα και άναρχη Μάλιστα, εδώ, ακριβώς επειδή έχει κυρωθεί η Διεθνή Συμφωνία για την παράτυπη εργασία και επειδή υπάρχουν και άλλες συμφωνίες οι οποίες θα κυρωθούν πριν το 23-24 βλέπουμε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Βιετνάμ είναι προκλήσεις που οφείλονται στις υπερβολικές δυνατότητες ε, και δραστηριότητες αλληλείας, ε, στην ε, υπεραλίευση και χρειάζεται παρακολούθηση εδώ από μέρους της Επιτροπής και στήριξη όταν επιτυγχάνεται πρόοδος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό να έχουμε μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης. Αυτή η εμπορική συμφωνία, αυτή η συμφωνία για αύξηση των επενδύσεων στην περιοχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και κάποιες άλλες πτυχές όπως την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, τη βιωσιμότητα και με αυτές τις εμπορικές συμφωνίες έχουμε τη δυνατότητα, διαθέτουμε ένα εργαλείο να ασκήσουμε πίεση στο Βιετνάμ έτσι ώστε να υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές ε, αλίας, να καταπολεμήσει την παράνομη και λαθρέα και άναρχη αλία, να υιοθετήσει αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής νομοθεσίας. Πιστεύω ότι έχουν καθοριστεί κάποιοι δασμοί, κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί είτε μερικώς είτε εντελώς, αυτή η συμφωνία μας δίνει τη δυνατότητα μιας πιο μεγάλης μεταβατικής περίοδου, έτσι ώστε οι τοπικοί παράγοντες να προλάβουν να υιοθετήσουν κάποιες από αυτές τις νέες προδιαγραφές. Επίσης, η συμφωνία τους επιτρέπει να λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο, εάν δούμε ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις επί της τοπικής παραγωγής λόγω της αύξησης των ε, εισαγωγών. Το θέμα της κίτρινης κάρτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία η οποία θα πρέπει να την εξετάσουμε και εκτός αυτής της συμφωνίας. Ε, το θέμα είναι να λαμβάνονται τα σωστά μέτρα, να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτηρεί, να παρακολουθεί αυτά που κάνει το Βιετνάμ και όλα τα κράτη-μέλη σε όλους τους τομείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πολλές ευκαιρίες. Πρόκειται για μια τεράστια αγορά, 95 εκατομμύρια κάτοικοι και πέρα από τα εμπορικά αυτά ωφέλη, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να έχει σαν σκοπό τη βελτίωση της ε, κατάστασης στη χώρα αυτή και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Παγκαθαουρούτουα. Κοιτάξτε, όπως και εσείς είπατε, πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία, η αλληλευτική συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως ευχαριστούμε τον κύριο Μπαρτόλο και υποστηρίζουμε πολύ την εργασία του. Ε, στις ε, τροπολογίες που θα υποβάλουμε θα προσπαθήσουμε να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο ε, την γνωμοδότηση έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τρία-τέσσερα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία ανέφερε η προελίσσα σας συνάδελφος. Ε, η κίτρινη κάρτα, πολύ σημαντικό ε, στοιχείο, καθώς επίσης ε, και οι ελλείψεις στα συστήματα ελέγχου είναι δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε και μέσω της, τροπολογίας που θα υποβάλουμε να ενδυναμώσουμε, να εντείνουμε. Πρώτον γιατί αφορά την βιωσιμότητα που είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στίχημα μεγάλο. Και δεύτερον, θέλουμε να ενδυναμώσουμε επίσης ε, το θέμα των εργασιακών παραβιάσεων, δηλαδή παραβιάσεων της εργασιακής ε, ε, νομοθεσίας για τους εργαζόμενους στον τομέα της αλίας, άλλωστε και παράβαση των συμφωνιών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Εάν η έλεγχη στο Βιετνάμ δεν μπορεί να είναι αρκετά σαφή και αποτελεσματική, ε, τότε θα φτάσουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα τα οποία ε, και θα δημιουργήσουν πρόβλημα ε, λόγω της εστρέβλωσης ε, του ανταγωνισμού και λόγω της παραβίασης ευρωπαϊκών διεθνών συμφωνιών. Γι' αυτό, γι αυτό ακριβώς αξιολογούμε πολύ θετικά την εργασία του εισηγητού, τον εμπιστευόμαστε, αλλά θέλουμε να τον βοηθήσουμε έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο δυνατή αυτή η γνωμοδότηση, να χρησιμοποιήσει δηλαδή τους όρους αυτούς που η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει σαν βασικά στοιχεία κλειδιά και τις, ε, είναι αρχές που τις συμμεριζόμαστε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπαρτόλο για τη δουλειά που έχετε κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αναφερθήκατε σε τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι έχουν ε, ε, φτάσει στα χέρια μας. Η προθεσμία υποβολής είναι αύριο. κυρία Σάλιβαν. Η κυρία Κόντε, ε, ένας από τους λίγους ε, στόχους που έβαλε στην επιστολή της ε, η κυρία Βάντερ Λάγεν ήταν ακριβώς η καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Τώρα βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ που έχει ήδη πάρει κίτρινη κάρτα για την παράνομη αλεία. Εάν πραγματικά βελτιώνονται οι συνθήκες σε μια χώρα μέσα από αυτές τις συμφωνίες, και αυτό ισχύει όντω, δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα και προκλήσεις. Στη δέκατη θέση είχε βάλει η αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία το, τα ψάρια τα οποία προέρχονται από το Βιετνάμ λόγω ακριβώς των βαρέων μετάλλων. Ε, εμείς δίνουμε όμως 15 δις ευρώ ε, και εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι γίνονται σεβαστές οι απαραίτητες συνθήκες τότε θα φτάσει στο τραπέζι μας ε, ψάρι το οποίο θα είναι πολύ κακής ε, ποιότητος. Ε, και επίσης υπάρχει, διατρέχουμε τον κίνδυνο να προέρχονται τα ψάρια αυτά από παράνομη αλία. Δεν είναι δυνατόν επίσης να παίζουμε και με την παράνομη αλία και με την αλία που δεν σέβεται τους υγειονομικούς κανόνες. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτόνομη όσον αφορά την αλία και επομένως η εμπορικές συμφωνίες είναι απαραίτητες. Ωστόσο, ε, δεν ε, είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Μπορούμε να ε, ε, χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους ε, ε, πόρους, τα όσα μας δίνουν οι θάλασσές μας, όχι μέσω υπεραλίευσης, με άλλους τρόπους. Υπάρχουν ψάρια τα οποία δεν τα καταναλώνουμε γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να τα καταναλώνουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας ή ότι δεν μπορούμε να εξάγουμε πλέον αυτά τα είδη ψαριών έτσι ώστε να έχουμε ε, ικανοποιητικά ε, αποτελέσματα. Ε, χαιρετίζω την εργασία του συναδέλφου Μπαρτόλο και τον του ζητώ να υποστηρίξει μέτρα καινούρια και καινοτόμες ιδέες μέσα στα πλαίσια αυτών των ήδη από καιρό υφισταμένων συμφωνιών. Πρέπει οπωσδήποτε οι ευρωπαϊκοί πόροι, οι ιταλικοί πόροι ή οι πόροι που προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος θα πρέπει να αξιολογηθούν πολύ περισσότερα και να προωθηθούν με εντονότερο ρυθμό. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ε, ομιλητής. Του Ο κύριος Γκονσάλες Κασάρες. Ε, ε, αυτό το ζήτημα σχετικά με την κίτρινη κάρτα του Βιετνάμ βεβαίως ε, είναι προβληματικό και μας ε, απασχολεί. Έχουμε τροπολογίες πάνω σε θέματα τα οποία μας απασχολούν, όπως ας πούμε αυτά τα 11.500 τόνοι τόνου που θα εισαχθούν. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό. Επίσης, κονσέρβες ε, τόνου καθώς επίσης ε, και οι αντίστοιχοι ε, δασμοί. Είναι σημαντικό θέμα αυτό. Εμείς δεν ε, είμαστε αντίθετοι με αυτήν την συμφωνία, ε, όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε απαιτήσει ε, οι οποίες είναι απαραίτητες, καθώς επίσης και θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. And Mr. Και ο κύριος Μιγιανμόν. Η περίπτωση του Βιετνάμ είναι από αυτές τις περιπτώσεις ε, που, ε, που υποδεικνύει γιατί η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡ και η Γενική Διεύθυνση Trade θα πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα. Ε, γιατί από τη μία μεριά έχουμε την παράνομη αλλήλεια και την ανεξέλεγκτη και από την άλλη μεριά διαπραγματευόμαστε εμπορικές συμφωνίες όπου αυτά τα σημεία δεν αναφέρονται ιδιαίτερως. Σε πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι, θα πρέπει να συντονίσει καλύτερα τα εμπορικά της προγράμματα και τα θαλάσσια ε, προγράμματα γιατί οι ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με χώρες οι οποίες αποδεδειγμένα ε, δημιουργούν προβλήματα, αυτό είναι λίγο παράλογο. Από τη μία μεριά δηλαδή ε, τους απειλούμε με κλείσιμο των εξαγωγών ε, και από την άλλη μεριά ανοίγουμε την ευρωπαϊκή αγορά σε όλα τα λευτικά προϊόντα που έρχονται από το Βιετνάμ. Αυτό είναι αντιφατικό και ε, αποτελεί έτσι μία κοντραντίξιο in Οπωσδήποτε λοιπόν οι πολιτικές θα πρέπει να είναι ε, πιο συντονισμένες έτσι ώστε να έχουν και καλύτερο αποτέλεσμα. Τούτου λεχθέντος ε, σε σχέση με το Βιετνάμ και άλλες ε, ασιατικές χώρες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την αλληλεία. Πρόκειται για χώρες οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερως ή μάλλον στις οποίες υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η παράνομη αλληλεία και εδώ μιλάμε για 12.000 τόνους Ε, η Ταϊλάνδη είναι η μεγαλύτερη παραγωγός ε, κονσερβών τόνου ε, και εάν ας πούμε απελευθερώνουμε τους δασμούς για την Ταϊλάνδη τότε θα κατεστρέφεται η βιομηχανία του, του τόνου και στην Ισπανία και αλλού. Εν πάση περιπτώσει Έχουμε μπροστά μας και τις διαπραγματεύσεις ε, με την ε, Ταϊλάνδη ε, και γι' αυτό θέλω να πω στην Κομισιόν ότι τα αλλιευτικά προϊόντα θα πρέπει σε όλες αυτές τις χώρες να θεωρηθούν ευαίσθητα, όχι μονάχα στο Βιετνάμ και εδώ δράτουμε της ευκαιρίας ε, ακριβώς για να πω ότι ε, ε, έχουμε σε λίγο μπροστά μας την συμφωνία με την Ταϊλάνδη. Γι' αυτό λοιπόν να μην καταστρέψουμε με την ανάστροφη του χεριού και με μία κίνηση την ευρωπαϊκή βιομηχανία, μεταποιητική βιομηχανία. So, over Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Κομισιόν, ακούσατε από όλα τα μέλη, από τους εισηγητές, την, ε, τον προβληματισμό τους. Ε, οι διερμηνείς δεν ακούν. Έκλεισε το μικρόφωνο του Προέδρου. Έδινε το λόγο στην Κομισιόν. Έλεγα λοιπόν ότι ακούσατε τους εισηγητές, ακούσατε ε, τον προβληματισμό των μελών για αυτή τη διαδικασία κίτρινης κάρτας, για τους ελέγχους. Να μας πείτε εάν ε, ε, πραγματικά πρέπει να αντιδρούμε κάθε φορά. Ο κύριος Μιγιανμόν ε, είπε ότι η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και η Γενική Διεύθυνση Τρέντ θα πρέπει οπωσδήποτε να συντονίζονται, να συνεργάζονται περισσότερο. Έχουμε την κυρία Γκαρσία από την Τρέντ και τον κύριο Νούνσα από την DG ΜΑΡΕ. Πέστε μας λοιπόν ό,τι έχετε στην ψυχή σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και τον συντάκτη της γνωμοδότησης και τους ευρωβουλευτές για τις επικοτομητικές παρατηρήσεις τους. Όσον αφορά την αντιπροσωπεία της ΣΥΝΤΑ που πήγε στο Βιετνάμ πριν από δύο εβδομάδες, πήγαν εκεί πέρα για να αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και συμφωνία προστασίας των επενδύσεων που συνάπτεται με το Βιετνάμ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Οι συνάδελφοι από την ντα λοιπόν επέστρεψαν με πολύ θετικέ αντιπώσεις θεωρούν ότι η κυβέρνηση του Βιετνάμ πραγματικά θέλει να σημειώσει πρόοδο σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία έχει θίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι όχι μόνο στο ζήτημα τη Αλλεία και δι τη καταπολέμηση παράνομη αδήλωτη και ανεξέλεκτη αλεία, αλλά και σε όλα τα περιβαλλοντικά αλλά και εμπορικά ζητήματα. Έχουμε μια πραγματική δέσμευση και προσήλωση από πλευρά του Βιετνάμ προκειμένου να σημειωθεί πρόοδο και να καταφέρουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Να σα υπενθυμίσω ότι πέρυσι πήγε και η δική σα όμω Επιτροπή στο Βιετνάμ, μια ομάδα ευρωβουλευτών λοιπόν είχε τη δυνατότητα εκεί πέρα να συνομιλήσει με τις βιετναμέζικες αρχές κάναν συγκεκριμένε επισκέψει και έμειναν πολύ ικανοποιημένοι, αν θυμάμαι καλά, από την επίσκεψη αυτή. Δείτε το δελτίο τύπου, το οποίο εξέδωσαν οι ευρωβουλευτέ, ε, καθότι πολλοί από του ευρωβουλευτέ που μετέβησαν τότε στο Βιετνάμ δεν συμμετέχουν στο νέο κοινοβούλιο. Πάντω έγινε μια αξιολόγηση ήδη από την Επιτροπή Αλία πέρυσι όσον αφορά το Βιετνάμ τώρα. Όσον αφορά τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη συμφωνία αυτή. Στα πλαίσια τη συμφωνία Δεύτερων Συναλλαγών υπάρχει ένα κεφάλαιο εμπορίου και βιώσιμη ανάπτυξη, προσπαθούν να καλύψουμε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική, περιβαλλοντική και εργατική πτυχή. Έχουμε εκεί ένα κεφάλαιο για την αλληλεία όπου αναφερόμαστε στη βιωσιμότητα των ελευτικών πόρων και τη υδατοκαλλιέργεια και οι δύο πλευρέ θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα διεθνή εργαλεία και να συνάδουν με τους διεθνείς κανόνες. Έχουμε επίσης μια συμφωνία για την καταπολέμηση της παράνομης αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλίας και εκεί έχουμε και την κίτρινη κάρτα η διαδικασία όμως FTA και η διαδικασία της κίτρινης κάρτας είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες που όμως είναι αλληλένδετες παράλληλα. Όσον αφορά τον συντονισμό, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πολύ καλός συντονισμός μεταξύ της DigiTrade και της DigiMaret. Η εμπορική συμφωνία συνήφθη το 2015. Έκτοτε είχαμε όλα αυτά τα διαδικαστικά βήματα, τη μετάφραση της συμφωνίας. Τον Οκτώβριο του 2017 είχαμε την κίτρινη κάρτα και έκτοτε είμαστε σε στενή επαφή με την DG Mare προκειμένου και οι δύο διαδικασίες να κινούνται παράλληλα. Πρόκειται για δύο πάντως ξεχωριστές διαδικασίες, αλληλένδετες βέβαια, και πιστεύω ή θέλω να ελπίσω ότι στα πλαίσια τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα μα δοθούν περισσότερε ευκαιρίε για να συζητάμε για τα ζητήματα αυτά με το Βιετνάμ. Τώρα, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργατικά δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα προφανώ ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα ευαίσθητο τομέα, αλλά θεωρώ ότι όντας περισσότεροι εμπλεκόμενοι πλέον με το Βιετνάμ στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Τώρα, όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, όπου υπάρχουν συγκεκριμένε δεσμεύσεις στα πλαίσια της συμφωνίας τέτοιων συναλλαγών, έχει σημειωθεί πρόοδος από το Βιετνάμ, για παράδειγμα. Μια βασική σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις έχει ήδη εγκριθεί από το Βιετνάμ και έχει δεσμευτεί το Βιετνάμ να καταπολεμήσει την κατανακαστική εργασία και επίσης έχει δεσμευτεί του χρόνου να προωθήσει όλη εκείνη την νομοθεσία που έχει να κάνει με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το Βιετνάμ προβαίνει σε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, ιδίω όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, όσον αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατά αυτόν τον τρόπο το Βιετνάμ ουσιαστικά προετοιμάζεται για την πολύ σημαντική αύξηση του εργατικού δυναμικού που θα έχει στο μέλλον. Η έγκριση λοιπόν τη συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα μα βοηθήσει να προωθήσουμε και να επιταχύνουμε όλε αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Επίσης, όσον αφορά την πρόσβαση αγορών, στα πλαίσια της FTA προσπαθούμε να απελευθερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερου τομεί. Αυτό έχει δεσμευτεί να κάνει και το Βιετνάμ. Τα πάντα θα, θα ελευθερωθούν μετά από την πάροδο 7 χρόνων. Εμεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι τομεί οι οποίοι είναι ευαίσθητοι. Για παράδειγμα, στα πλαίσια τη εμπορική ελευθέρωση δεν καλύπτεται ο τόνος σε κονσέρβα είναι ένας τομέας ο οποίος είναι αρκετά ευαίσθητος και αποφασίσαμε να τον αποκλείσουμε από τη συμφωνία για να μην δημιουργηθεί προηγούμενο. Έτσι λοιπόν όταν θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Ταϊλάνδη θα έχουμε πάλι μια περιορισμένη ποσόστοση όσον αφορά τον τόνο σε κονσέρβα, όπως ακριβώς κάνουμε τώρα δηλαδή με το Βιετνάμ. Εν κατακλείδη, ελπίζω ότι θα δώσετε εσείς μια θετική γνώμη για τη συμφωνία αυτή, η οποία θεωρούμε ότι θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές, για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, τους ε, καταναλωτές του Βιετνάμ, για τα εργατικά δικαιώματα και προσβλέπουμε ότι θα έχουμε μια θετική συνεργασία με εσάς. Σας ευχαριστώ. Κύριε δεν είναι εδώ. Είμαι η Εύα Πλέκραν και εργάζομαι στην Digimare όσον αφορά τη σχέση νομίζω με την ε, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, ο, η συνάδελφος νομίζω έδωσε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Συνεργαζόμαστε και αφού συναυθεί η συμφωνία, αλλά και κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων και βημάτων πρόοδου, συμμετέχουμε στη διαπραγμάτευση σε διάφορες ομάδες εργασίας, αυτή που ασχολάται με την βιωσιμότητα, την πρόσβαση στην αγορά, τη χρήση των ονομασιών προέλευσης κτλ. Ε, είμαστε λοιπόν σε συνεργασία μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων. Όλα ωραία και καλά. Δεν μας είπατε όμως πότε θα δώσετε πράσινη κάρτα στο Βιετνάμ. Μπορώ να σας απαντήσω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι μία ομάδα βρίσκεται στο Βιετνάμ, αξιολογεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης σίγουρα θα είναι σημαδιακό για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Βιετνάμ. Όλα αυτά θα βασιστούν σε ανάλυση και σε μία ε, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από εδώ και πέρα. Ωραία. Ναι, ναι, λέει ο πρόεδρος. Ναι, ε, μου λένε ότι αυτό μπορεί να πάρει τρία με πέντε χρόνια. Ξεκινήσαμε το 17 παρόλα αυτά. Ο εισηγητής. Συντάντο, ε... Κύριος Μπαρτόλο, ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ τις αμφιβολίες ε, για τους δισταγμούς ε, των ε, συναδέλφων. Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε και τα όσα κάνει το Βιετνάμ ε, επί τη βάση των στοιχείων που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπωσδήποτε η συμφωνία με το Βιετνάμ είναι συμφωνία που είναι καλό να ολοκληρωθεί. Ε, γιατί αν δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή, στην ουσία ε, θα έχουν αποβεί μάταιες οι προσπάθειες της χώρας ε, για βιωσιμότητα του αλλιευτικού τομέα και θα αφήνει απ' έξω έναν εταίρο, τον οποίο αμέσως θα έπαιρνε υπό την επιρροή της η Κίνα, ας πούμε, ή άλλες χώρες της γειτονιάς. Υπάρχουν ήδη, είναι γεγονός μεγάλες εισαγωγές από την ε, χώρα αυτή. Βεβαίως είμαστε έτοιμοι να ε, ενισχύσουμε τις ε, προϋποθέσεις απέναντι στο Βιετνάμ, να υποστηρίξουμε τις αμφιβολίες σας, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και πρέπει να δεχτούμε λοιπόν ότι η χώρα αυτή καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες και πιστεύω ότι και η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να εκφράσει θετική άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι αύριο στις 5. Και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπαρτόλο για την ε, συμβιβαστική σας διάταση, διάθεση. Και βεβαίως, αν υπάρξει ανάγκη για συμβιβαστικές τροπολογίες, να τα συζητήσετε μεταξύ σας και ε, θα, ψηφιστεί το, η ψηφοφορία θα γίνει στις 4 ε, Δεκεμβρίου. Επόμενο θέμα, η παράταση του πρωτοκόλου ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας όσον αφορά το πρωτόκολλο βιώσιμης για την Ελία και της εταιρικής σχέσης, συγγνώμη και της Συμφωνίας Σύμπραξης έχει ξεκινήσει η διαδικασία συνένεσης στο Συμβούλιο, ε, αλλά μπορώ αμέσως να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, εάν έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της Κομισιόν που θα είχε την διάθεση να μας μιλήσει για την Μαυριτανία. Καλή σας ημέρα. Το Συμβούλιο την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου ενέκρινε την παράταση του ε, ισχύοντος πρωτοκόλλου με την Μαυριτανία. Το ισχύον, το υφιστάμενο πρωτόκολλο, όπως γνωρίζετε, ε, έλυγε την 8η ε, Νοεμβρίου και στα πλαίσια της εντολής ε, που μας έδωσαν τον προηγούμενο Ιούλιο τα κράτη-μέλη, θεωρήθηκε ότι καλό θα ήταν, σημαντικό θα ήταν να παραταθεί για ένα χρόνο το πολύ ακόμα αυτό το πρωτόκολλο εν αναμονή της πραγματικής του ε, με Ανανέωση. Πρόκειται στην ουσία για ε, μια συμφωνία και ένα πρωτόκολλο και πρέπει οι διαπραγματεύσεις να γίνουν από κοινού. Μια και αναμένονται περίπλοκες διαπραγματεύσεις αυτές, τα κράτη-μέλη θεώρησαν ότι θα έπρεπε να παραταθεί για ένα χρόνο το ισχύον πρωτόκολλο. Ο πρώτος γύρος συζητήσεων έγινε το Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Μαυριτανία συμφώνησαν επί ενός κειμένου ανταλλαγής επιστολών που προβλέπει την παράταση του πρωτοκόλου για ένα χρόνο. Ε, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Σεπτεμβρίου όμως ήδη αρχίσαμε να συζητούμε το κείμενο της συμφωνίας και την προηγούμενη εβδομάδα ε, ε οργανώθηκε δεύτερος γύρος ε, ε, συζήτησης που αφορούσε πλέον και το πρωτόκολλο και τη συμφωνία. Επιστρέψαμε από την Μαυριτανία την, το προηγούμενο Σάββατο. αυτή τη βδομάδα προβλέπεται ε, η ε, υπογραφή έτσι ώστε να μην υπάρξει διακοπή των ε, ευρωπαϊκών αλλιευτικών ε, δραστηριοτήτων ε, στα είδη της Μαυριτανίας. Δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε για όλα με τη μία, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει ή εν πάση θα πρέπει να αποφευχθεί η εν θα πρεπει να αποφευχθει η διακοπη ε, των δραστηριοτήτων. Τον Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες προβλέπεται ο επόμενος γύρος και ευελπιστούμε ότι για το πρωτόκολλο και τη συμφωνία τον, την άνοιξη του 2020 να έχουμε ολοκληρώσει έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, οποιαδήποτε ε, διακοπή το Νοέμβριο του 2020. Δηλαδή μέχρι τότε να έχει τεθεί σε ισχύ και το πρωτόκολλο και η συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σχόλια, ερωτήσεις, θέλετε κάτι να πείτε. Ε, Κύριε Πρόεδρε, μια σύντομη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την κατάρτιση ζωνών. Έχετε καταλήξει κάποια συμφωνία με τις ζώνες αυτές, οι οποίες θα πρέπει να φτάνουν και κοντά στην παράκτια περιοχή, προκειμένου οι τοπικές κοινότητες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αλλιευτικά αποθέματα τα οποία βρίσκονται κοντά στις ακτές και θα μπορούσατε να μας δώσετε επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των παρακτήων ζωνών. Δεν νομίζω θέλει να πάρει κανείς άλλο το λόγο. Ο κύριος Μιλάν παρακαλώ. Ε, κοιτάξτε, είναι όντως πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία. Ε, όμως ε, η μέθοδος αυτή της ε, παράτασης για ένα χρόνο έτσι ώστε να μην υπάρξει διακοπή όσον αφορά την παρουσία του Ευρωπαϊκού Στόλου. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω το πρόβλημα που έχουμε στο βόρειο σύνορο της Μαυριτανίας, ε, στα όρια λοιπόν του, του, του Βορρά, ε, που μπλοκάρουν ε, φορτηγά ψυγεία με φρέσκα ψάρια θα πρέπει να βρεθεί... Ναι, ξέρω ότι υπάρχει αυτή η ειδική κατεξαίρεση διαδικασία ε, που επιτρέπει στα πλοία να φτάσουν στο Ουαντιμπούλ και όχι στην Τάχλα, αλλά θα πρέπει να δούμε εάν αυτή ε, η ειδική διαδικασία λειτουργήσει. Το πρόβλημα είναι ότι ε, πολλές φορές έχουμε επιθέσεις κατά αυτών των κονβόι των φορτηγών που πολύ συχνά είναι ισπανικά φορτηγά. Η κατάσταση είναι ε, περίπλοκη. Τώρα, εάν με αυτές τις ειδικέ ασκήσεις κατά κάποιο τρόπο καταφέρουμε να ξεμπλέξουμε μία περίπλοκη κατάσταση, τόσο το καλύτερο. Ωστόσο, ε, αυτός ο μηχανισμός ίσως θα πρέπει να καθιερωθεί στη νέα συμφωνία γιατί ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις εκφορτώσεις ε, και, στο, και τις εκφορτώσεις του Γουαδιμπού. Ευχαριστώ. Επιτροπή, μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ναι, όσον αφορά τις διάφορες ζώνες αλίας, όπως σας είπα, το πρωτόκολλο επεκτείνει τις ίδιες ακριβώς ε, προδιαγραφές. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα όσον αφορά τις ζώνες αλίας, όπως είχαν καθοριστεί με σκοπό να μπορεί να δραστηριοποιηθεί ο τοπικός αλλιευτικός στόλος. Δεν υπάρχει λοιπόν επαναλαμβάνω τροποποίηση με αυτό το νέο πρωτόκολλο. Όσον αφορά τώρα το σύστημα και τις δυσκολίες που όντως αντιμετώπισαν κάποια φορτηγά που βρισκόταν στα σύνορα Μαρόκου Μαυριτανίας. Δυσκολίες που ουσιαστικά δίναν τη δυνατότητα σε κάποια σκάφη να εγκαταλείψουν τα λιμάνια αυτά, να μπορέσουν να μπουν σε, στα κοντινότερα λιμάνια στο Μαρόκο. Από ό,τι φαίνεται η συνεργασία με τις αρχές Μαυριτανίας ήταν εξαιρετικές, τέλειες και τελικά δεν χρειάστηκε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διότι τα ε, οχήματα αυτά απελευθερώθηκαν και μπόρεσαν να περάσουν από τα σύνορα. Αλλά είδαμε ότι στην ε, θεωρία τουλάχιστον το εναλλακτικό αυτό σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει με ευελιξία. Αυτό αποτελεί μάλιστα και αντικείμενο των διαπραγματεύσεων που εκκρεμούν. Η πρώτη μεικτή επιτροπή θα συνεδριάσει το Δεκέμβριο παράλληλα με τις άλλες διαπραγματεύσεις και θα κάνει ένα ε, απολογισμό αυτής της επιτυχημένης μέχρι τώρα διαδικασίας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή μπορούμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα να πούμε ότι την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε θα γίνει η παρουσίαση της έκθεσης. νεγάλη είναι το επόμενο θέμα και αυτή τη στιγμή περιμένουμε την σύμφωνη γνώμη. Το θέμα αυτό το έχει αναλάβει η ομάδα Renew Europe. Κύριε Μπέργκ, εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να σας παρακολουσιάσω αυτό το νέο πρωτόκολλο που πρόσφατα έχει μονογραφηθεί Πρόκειται για μια συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια πριν το 2000, διεκόπη το 2000 και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε με την χώρα αυτή διαπραγματεύσεις και συμφωνίες καθότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική χώρα. Η Αλία παίζει καθοριστικό ε, ρόλο και αυτά που συμβαίνουν στα ύδατα της Σενεγάλης επηρεάζουν και όλες τις ε, γύρω περιοχές. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει εταιρική ε, σχέση, ένας σημαντικός παράγοντας για τη Δυτική Αφρική. Μετά από την πρώτη σειρά διαπραγματεύσεων συμφωνήσαμε με τη Σενεγάλη και υπάρχει, όπως σας είπα, από τις 19 Ιουλίου η πρώτη συμφωνία εξαιρετική συνεργασία πρέπει να σας πω με τις αρχές της Σενεγάλης και πρόκειται για μια συμφωνία η οποία συμπεριλαμβάνει αν θέλετε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 25 άτομα συμμετείχαν σε αυτές τις ε, διαβουλεύσεις και συζητήσεις. Το σύνολο λοιπόν του τομέα της Αλίας είχε εκπροσωπηθεί και εκπροσωπήθηκε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για μια συμφωνία με διάρκεια πέντε ετών. Αυτό είναι κάτι θετικό για μένα, για να υπάρχει σταθερότητα όσον αφορά τα ωφέλη, τα έσοδα για τη χώρα αυτή. Δυνατότητες αλίας για τα, τις μηχανότρατες, 28 ε, θυναλιευτικά, 10 λιευτικά με καλάμι, 5 παραγαδάρικα και όπως σας είπα και 2 μηχανότρατες. Ε, κάτι το οποίο επιτρέπει και στον ε, αλλιευτικό στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν σε αυτήν την ε, εμπειρική θα έλεγα αλία. Όσον αφορά το 1.700.000 που είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το χρόνο, 900.000 είναι η συμμετοχή στην δραστηριοποίηση του τομέα. Στηρίζουμε δηλαδή τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλίας, τη Σενεγάλη, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη στήριξη στην αλλία μικρής κλίμακας και την ερευνητική δραστηριότητα. Επιμένω αυτό γιατί είχαν προγραμματιστεί κάποια επιστημονικά προγράμματα τα οποία δεν είχαν χρηματοδότηση και δεν προχώρησαν ε, τα προηγούμενα χρόνια. Με το νέο αυτό πρωτόκολλο μπορούμε να στηρίξουμε όλη την ερευνητική δραστηριότητα σε Νεγάλη. Συμμετοχή των πλειοκτήτων, επίσης, με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία. Αν βάλουμε λοιπόν από κοινού τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή των πλειοκτητών, ξεπερνάμε τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα χρηματοδοτήσουν την Σενεγάλη στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Τώρα, όσον αφορά τις ε, ε, ποσότητες, έχουμε τον τόνο και το μπακαλιάρο, το είδος ε, αυτό της Σενεγάλης. 14.000 τόνους, 10.000 τόνους. 2.000 τόνοι μειώνεται σε 1.750 1.750 τόνους. Οι ποσότητες εδώ μειώνονται στα πιο ευάλωτα αποθέματα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει παρακολούθηση αυτής της αλληλευτικής δραστηριότητας. Έχουμε παρατηρητές ε, πάνω στα σκάφη με δυνατότητες ε, επίσης περίοδων διακοπής. Τεχνικά μέτρα τα οποία έχουν ε, βελτιώσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης, για να αποφευθεί η αλία θηλαστικών, θαλάσσιων θηλαστικών και πτηνών. Πρόκειται λοιπόν για μια συμφωνία η οποία θεωρούμε ότι θα έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθώς και το σεβασμό του οικοσυστήματος και του θαλάσσιου περιβάλλοντος στα ύδατα της Σενεγάλης. Ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτήν την συμφωνία και αυτήν την ανανέωση της εταιρικής σχέσης μας με τη Σενεγάλη. Ευχαριστούμε και εμείς ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Μία ερώτηση έχετε. Ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να υποστηρίξω αυτή τη σημαντική συμφωνία. Είναι σημαντική για τον ελληνικό τομέα της Ευρώπης, της Ισπανίας και της χώρας των Βάσκων. Ευχαριστώ την Κομισιόν ε, για τις προσπάθειες τις οποίες έχει καταβάλει, γιατί έχουν ε, ε, υπάρξει πολλές περιπλοκές. Βλέπουμε επίσης και αύξηση της συμβολής των πλειοκτητών ε, και την ε, ε, ευαισθησία όσον αφορά την ανάπτυξη του τομέα. Η ανάπτυξη του τομέα για και λόγω των επιστημονικών λόγων που ευθυγραμμίζονται και με τις κεντρικές γραμμές της Συμφωνίας Σύμπραξης. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου, λέει ο κύριος Γκονζάλης Κασάρες, ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η συμφωνία και για την Ισπανική και για την Γαλλική, ε, ε, για το Γαλλικό στόλο και για το στόλο της Γαλλικίας. Θα πρέπει να έχουμε πραγματικά, να κάνουμε μια συμφωνία όπως ε, υπόθηκε και προηγουμένως, έχουμε και παραγαδιάρικα, έχουμε και ε, θυναλιευτικά με καλάμι, έχουμε και ε, μηχανότρατες και επομένως όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και μηχανότρατες επίσης. Το οικονομικό ποσό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, ενδιαφέρουν όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Νομίζω ότι και για την τρίτη χώρα ε, είναι πάρα πολύ σημαντική ε, και νομίζω ότι είναι καλό να κάνουμε μια τέτοια συμφωνία η οποία θα είναι επωφελής προς όλους. Ευχαριστούμε. Δεν νομίζω ότι τέθησαν συγκεκριμένε ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι δεν είναι. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Έχουμε παρεμπίπτους αλλοί όσον αφορά τον μπακαλιάρο της Συνεγάλης ή όσον αφορά την αλίευση του τόνου. Υπάρχουν και πέρα συγκεκριμένοι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να τηρηθούν. Αυτή είναι η ερώτηση που σας θέτω εγώ. Και μια σύντομη απάντηση περιμένουμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει κάποια παρεπίπτουσα σίγουρα, αλλά πάντα σε αποδεκτά επίπεδα η αλία της Σενεγάλης δεν διαφέρει πάρα πολύ από την αλία στις όμορες χώρες. Σαφώς υπάρχει παρεπίπτους αλία, η οποία όμως θα πρέπει να δηλώνεται κάθε φορά. Αυτό είναι ένας γενικός ο οποίος ισχύει και σε κάθε περίπτωση τα δηλωθέντα τουλάχιστον ε, ποσά είναι αποδεκτά και κυρίως όσον αφορά τον μπακαλιάρο της Σενεγάλης, και όσον αφορά την αλεία του από τις μηχανότρατες. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μπορούμε να έχουμε μια πιο συστηματική παρακολούθηση των αλευμάτων αυτών και όπως σας είπα αυτή τη στιγμή μέσω του πρωτοκόλλου αυτού δίνουμε τα παρέτα κίνητρα προς τη Σενεγάλη προκειμένου να μειώσει την του αλεία... τόσο ηχθειών όσο και θαλάσσιων θηλαστικών. Πρόκειται για κάποιες νέες διατάξεις οι οποίες θα έχουν ως στόχο να μειώσουν αυτού του είδους τα λιεύματα. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Και βέβαια περιμένουμε να μας προτείνετε και ένα χρονοδιάγραμμα όσον αφορά, για να εγκρίνουμε και εμείς την έκθεσή μας. Σας περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το περιθμό 21 πρόταση για την τροποποίηση του πρωτοκόλου της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των θηνοειδών του Ατλαντικού. Στην ομάδα ID κατενεμήθη σήμερα η έκθεση αυτή, δεν έχουμε ακόμα εισηγητή. Η κυρία Χάφορτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο, τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ σημειώσεις μου. Δεν φαίνεται να υπάρχει κυρία Χάφορτ αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, έτσι δεν είναι. Κάποιο άλλο, τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, έστειλα ε, ένα μήνυμα στη συναδελφό μου, αλλά φτάσατε πολύ νωρίτερα στο σημείο αυτό από ό,τι περιμέναμε. Νομίζω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα η συνάδελφος και δεν μπορώ εγώ να σας ενημερώσω για την ICAT, πάντως έχω στείλει ένα μήνυμα. μπορούμε να έχουμε την παρουσίαση αυτή στην επόμενη συνεδρίασή μας. Άλλωστε θα πάμε συνεδρίαση της ΆΙΚΑ το εξ ημών την επόμενη εβδομάδα. Και νομίζω ότι άλλωστε τα στοιχεία τα οποία μας δώσετε μιλάνε από μόνα τους σε σχέση με τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν σε Σύμβαση ICAT. Επομένως δεν θα καλύψουμε σήμερα το σημείο αυτό και δεν νομίζω ότι χρειάζεται γενικά τέτοιο λέει ο Πρόεδρος. Επομένως να στείλω ένα άλλο μήνυμα τώρα στην αδελφό μου. Μα, τι ωραία, γι' αυτό έχουμε και τα κινητά τηλέφωνα. Λοιπόν, δεν έχω παρά να σας πω αυτή τη στιγμή ότι οι συστάσεις των συντονιστών που εγκρίθηκαν σήμερα το πρωί σας έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ζητάμε να υποβάλλετε αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις όταν θα έχετε το χρόνο να διαβάσετε τα πρακτικά αυτή. Αυτά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Στα διάφορα έχουμε κάποιο άλλο ζήτημα, όχι. Επομένω, βλέπω ότι είναι 5 και 25 και μόνο ότι κάναμε και 10 λεπτό διάλειμμα καταφέραμε να ολοκληρώσουμε εγκαίρω την ε, σημερινή συνεδρίαση.